Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Hay algunos miembros que... Καλημέρα. Κάποιοι δεν έχουν έρθει ακόμα, αλλά επειδή η μερίσια διάταξη είναι πολύ φορτωμένη, ας αρχίσουμε, αν μη τι άλλο, με τα προκαταρτικά. Στην ημερήσια ε, διάταξη έχετε δει τι περιλαμβάνεται, την έχετε στους φακέλους σας. Υπάρχουν αντιρρήσεις, Εγκρίνεται. Ελπίζω επίσης να διαβάσετε και τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων και πάλι αν δεν υπάρχει αντίρρηση θεωρούνται εγκεκριμένα. Τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων. Έχω διάφορες ανακοινώσεις να σας κάνω, αλλά επειδή έχουμε εδώ τους συναδέρφους από την Επιτροπή Ίντα και κυρίως τον κύριο Λάγκε, που και αυτός έχει και άλλες δουλειές σήμερα το πρωί, θα περάσουμε κατευθείαν την ε, κοινή ακρόαση που έχουμε οργανώσει για σήμερα το πρωί, οι δύο επιτροπές. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον για πάρα πολλούς από εσά και για πάρα πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για εμπειρογνώμονες και πολλούς που επέμειναν ότι έπρεπε να εξετάσουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις τεχνολογίες ψυχιακής παρακολούθησης και συστήματα παρεμβολής. Είναι ένα θέμα όλο ιδιαίτερος ενδιαφέρον για τα επόμενα χρόνια. Και τώρα, αλλά όσο περνά καιρός όλο και περισσότερο. Η κοινωνία των πολιτών συνειδητοποιεί πολλά πράγματα, ενδιαφέρεται όλο και περισσότερο για τις ψηφιακές αυτές τεχνολογίες που γνωρίζουμε, αλλά την ε, ύπαρξή τους εμείς γνωρίζουμε περισσότερο από πολλούς άλλους. Η χρήση τους μπορεί να πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από αυτήν. Είμαστε εδώ σήμερα για να αναλύσουμε το θέμα, να δούμε κατά πόσο αυτά τα συστήματα παρακολούθησης φτιάχνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς χρησιμοποιούνται σε διάφορες χώρες ακριβώς για να μπορούν να ελέγχουν τους πολίτες, τους διάφορες οργανώσεις που διαμαρτύρονται, αντιπολιτεύονται κτλ. Θέλουμε να δούμε λοιπόν πώς ελέγχεται αυτή η κατάσταση. Η βασική ιδέα είναι ότι το πρώτο τμήμα της ακρόασης αυτής γίνεται από την Προεδρία του κύριου Λάγκε, του Προέδρου της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Σε αυτό το πρώτο τμήμα του πρωινού θα συζητήσουμε τον έλεγχο των εξαγωγών. Και στο δεύτερο τμήμα της ακρόασης, όπου θα προεδρεύω εγώ, θα δούμε τις σχέσεις των συστημάτων αυτών με τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουμε και την συνάδελφο και συγγήτρια για το θέμα αυτό, την κυρία Μαρέτη Σχάκε. Θα, της... θα δώσω το λόγο πρώτα στον κύριο Πλάνκε και μετά στην κυρία Σχάκε, προκειμένου να μας παρουσιάσουν το πρώτο τμήμα της σημερινής μας συζήτηση. Κύριε Λάγκε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε να προεδρεύσετε του πρώτου τμήματος σίγουρα είναι η αρχή μιας μεγάλης φιλίας ανάμεσα στην Επιτροπή σας, την Επιτροπή Ίντα και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σένα Έλενα. Όντως, η Επιτροπή μας είναι υπεύθυνη για τα θέματα εξαγωγής ε, προϊόντων και πολύ επισταμμένο ήδη έχουμε συζητήσει το θέμα των προϊόντων της χρήσης σε ό,τι αφορά τα θέματα hardware μηχανημάτων και άλλων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν θετικά ή αρνητικά και δεδομένη της ε, ολοένα και εξελισσόμενης ψηφιοποίησης το θέμα του hardware, του software αλλά και το θέμα της γνώσης για την ψηφιοποίηση μπαίνει συνέχεια και πιο, όλο και πιο πολύ το επίκεντρο και σε ό,τι αφορά και τις εξαγωγές ε, προϊόντων της ε, χρήσης. Νομίζω ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να είμαστε υπεύθυνοι για αγαθά τα οποία εξαγάγονται από την Ένωση και τα οποία ενδεχομένως χρησιμοποιούνται για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σε ό,τι αφορά τέτοιο υλικό και λογισμικό hardware και software υπάρχει αυτή η η αμφισημία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς αρνητικούς σκοπούς, αλλά και για να αγγίθουν για παράδειγμα, την ελευθερία, όπως έγινε στην Αραβική Άνοιξη, για προστατευτισμό, αλλά και για διευκόλυνση του εμπορίου. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για προπαγάνδα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για ενίσχυση της τεχνογνωσίας, για την παρακολούθηση, αλλά και για νόμιμα μέτρα ασφάλειας για βιομηχανική παρακολούθηση αλλά και για την ε, τήρηση και την διαφύλαξη των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι πολύ αμφίσιμη λοιπόν η δυνατότητα χρήσης αυτό του νέου ψηφιακού λογισμικού του υλικού και της σχετικής γνώσης. Γι' αυτό λοιπόν στο πρώτο επίπεδο το θέμα είναι οι εξαγωγές των άγαθων να συμφωνήσουμε επί κάποιων αρχών σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές και πρώτα δώσουμε το λόγο στους εμπειρογνώμονες, θα ήθελα να δώσω το λόγο καταρχάς στην εισηγήτριά μας, την κυρία Σκάκε. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καλωσορίζω όλους αυτή την κοινή ε, ακρόαση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο συμπροέδρους ε, οι οποίοι είναι αμφιτρίωνες ε, αυτού του, αυτής της εκδήλωσης γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική η αντιμετώπιση του θέματος και από πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και από πλευράς εμπορίου και είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες. Από το 2009 θα δούμε πώς έχουν εξελιχθεί και πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει αντίκτυπο στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, εμείς ε, εργαζόμαστε εδώ σε θέματα ε, τα οποία θα αντιμετωπιστούν σήμερα και από τους ομιλητές. Επίσης, Νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε μάλιστα τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από την προώθηση των τεχνολογιών, του, των τηλεπικοινωνιών, του διαδικτύου, ε, είναι στοιχεία τα οποία επιτρέπουν την γρήγορη ε, πρόσβαση ε, και δίνουν δύναμη στους πολίτες να ενημερωθούν εν ώψη εκλογών. Είναι ε, σημαντικό να έχουν οι πολίτες πρόσβαση σε αυτήν την τεχνολογία. Δεν πρέπει να λησμονούμε λοιπόν ότι οι τεχνολογίες έχουν βοηθήσει την πρόθεση και ανάπτυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αυτό δεν μπορεί να το αγνοήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, επίσης ε, θα πρέπει να δούμε τους κινδύνους που μπορούν, που μπορούν να υπάρξουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα εάν δεν χρησιμοποιηθούν ή αν χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα οι ευφυείς ε Είχαμε την Αραβική Άνοιξη πρόσφατα και άλλες εξεγέρσεις ε, οι οποίες χρησιμοποίησαν από τη μία πλευρά πολύ τις ε, τεχνολογίες και από την άλλη χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις περιπτώσεις οι τεχνολογίες ε, για παρεμβάσεις, καταστολές και παρεμβολές. Ε, ε, πολύ συχνά ε, η ανάπτυξη τεχνολογίας της, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις Ηνωμένε Πολιτείες είχαμε ανάπτυξη τεχνολογιών οι οποίες όμως μεταφερόμενες σε, σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν ε, να επηρεάσουν αρνητικά ε, εξελίξεις. Δηλαδή μπορεί να είναι ε, πολύ αρνητικές και για τα ανθρώπινα δικαιώματα εάν αυτού του είδους οι προηγμένες τεχνολογίες πέσουν σε λάθος χέρια. Από την άλλη πλευρά βεβαίως δεν είναι σωστό να πούμε ότι το θέμα αυτό αφορά μονάχα τις τρίτες χώρες και ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα παρεμβολών ή παρακολούθησης ή χρήσης τεχνολογίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τα δούμε όλα αυτά. Ε, η Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης ε, και στην ε, κλοπή βιομηχανικών μυστικών. Αυτό δεν μπορεί και δεν θα πρέπει, αν θέλετε τη γνώμη μου, να γίνεται μέσω χρήσης ενωσιακού υλικού. Είναι λοιπόν σήμερα μια ευκαιρία να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και τις επικαιροποιημένες πληροφορίες για όλα αυτά τα θέματα. Ε, εμείς στο δικό μας ψήφισμα λέμε ότι θα πρέπει να εντάξουμε τον ρόλο της τεχνολογίας χωρίς ε, ε, όμως ε, να επιβάλλουμε επιπλέον βάρος σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα πρέπει να αποφύγουμε στρατηγικούς κινδύνους και έχουμε ήδη αναγνωρίσει την ανάγκη να υπάρξει έλεγχος των εξαγωγών μέσω των τεχνολογιών. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο και επομένως εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι όσον αφορά τον κανονισμό για την ε, χρήση. Ε, υπάρχουν και άλλες πολιτικέ, ε, πολιτικές ε, οι οποίες δεν μπορούν να αποτρέψουν την νόμιμη χρήση της, της τεχνολογίας αλλά θα πρέπει να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι δημοσιογράφοι, ακτιβιστές κτλ να έχουν και αυτή πρόσβαση στην τεχνολογία της επικοινωνίας ας πούμε μέσω της αποκρυπτογράφησης ε, ε, ε, δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε ότι πλέον με το πάτημα ενός κουμπιού ή του ποντικού του υπολογιστή μπορεί να γίνει μεταφορά τεχνολογίας που μπορεί να έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο. Εμείς βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε αντιμέτωποι με την παγκοσμιοποίηση, με τον παγκόσμιο ιστό, με τις εξαγωγές. Θα πρέπει οπωσδήποτε να ενδυναμώσουμε και να τροποποιήσουμε τους κανόνες ε, που διέπουν το εξωτερικό μας ε, εμπόριο έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία αυτά. Είναι σημαντικό να εστιάσουμε την προσοχή μας ε, στο εμπορικό σκέλος της τεχνολογίας έτσι ώστε να αποφευθούν οποιαδήποτε παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω παρακολούθησης των εμπορικών συναλλαγών. Ποιος αγοράζει, τι αγοράζει, συστήματα παρεμβολή, συστήματα παρακολούθησης δεν θα πρέπει να δίνονται, να πολλούνται είτε σε ε, ε, ε, κυβερνήσεις είτε σε υπηρεσίες παρακολούθησης οι οποίες γνωρίζουμε ότι παραβιάζουν ανθρωπίνα δικαιώματα. Από την άλλη πλευρά βεβαίως οι εμπορικές συναλλαγές μπορεί να είναι νόμιμες αλλά ξέρουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, για ε, διάλυση συγκεντρώσεων ή ε, για την παρακολούθηση αντιφρονούντων κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε και τα στάνταρ της τεχνολογίας και τις προϋποθέσεις. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει καλύτερη ενσωμάτωση και συζήτηση και συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων έτσι ώστε να μην παίρνουν τις αποφάσεις ε, χωριστά ε, ε, για το εμπορικό σκέλος και για το σκέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπωσδήποτε θα πρέπει να ενσωματώσουμε και να σφυλατίσουμε μάλλον νέες συνεργασίες. Θα πρέπει οπωσδήποτε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να ενσωματωθεί στα εμπορικά ζητήματα έτσι ώστε να υπάρξει μια προστιθέμενη αξία και να προστατευτεί περισσότερο και η προσωπική ζωή ε, και όλες οι δραστηριότητες. Ε, αυτές ήταν οι αρχικές μου παρατηρήσεις. Ευελπιστώ ότι θα ακούσουμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα. Ε, είναι πολλά υποσχόμενο το πάνελ το οποίο έχουμε σήμερα μαζί μας. Ουσιώδου σημασία είναι να συμπεριλάβουμε στις διαδικασίες της ανάπτυξης ευθειών στρατηγικών να όλους αυτούς τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα θέματα και ευελπιστούμε λοιπόν ότι ακόμα περισσότερο θα αναπτύξουμε τις ενωσιακές ε, πολιτικές και όλο και περισσότερο θα εντάξουμε ε, την ανανέωση και τις νέες τεχνολογίες στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σάκη Έχουμε τώρα τρεις εμπειρογνώμονες στους οποίους ε, θα δώσω αμέσως το λόγο για 8 λεπτά στον καθένα και μετά θα ξεκινήσει ε, η διαδικασία των ερωτήσεων. Τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν ε, ερωτήσεις πολύ σύντομες ε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πρώτα απ' όλα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπένα Βάγνερ από το Πανεπιστήμιο της Λουμπλιάνα υπεύθυνο για το Κέντρο Διαδικτύου και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων the Duan Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εμπορικών Θέσεων που διοργανώνουν αυτή την ε, ε, συνάντηση και νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο, πολύ, τόσο πολλά άτομα, τόσο πολλοί όρθιοι εδώ πέρα στην αίθουσα καταδεικνύει πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην διαφάνεια αυτή βλέπετε πώς φτάσαμε εδώ, βλέπετε κάποιους διαδηλωτές έξω από μια Ιταλική εταιρεία γιατί ένας Ευρωπαϊκός Όμιλος είχε δώσει προϊόντα στην Συρία κατά τη διάρκεια των εξεργέσεων. Εδώ πέρα βλέπετε ότι αποκαλύφθηκε από τους δημοσιογράφους αυτό και οι κυβερνήσεις ε, δεν, δεν ήξεραν επακριβώς τι συνέβαινε. Χρειάστηκε δημοσιογράφοι να το αποκαλύψουν και βλέπετε εδώ λοιπόν ότι υπάρχουν στοχευμένα συστήματα παρατήρησης που χρησιμοποιούνται κατά των ακτιβιστών ε, στον κόσμο όλο και βλέπετε ότι είναι πάρα πολλά τα μέρη αυτά του κόσμου που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή και όπου αυτό ε, χρησιμοποιείται κατά των ε, ακτιβιστών. Οι διερμηνείς ε, και αυτοί οι άνθρωποι είναι. Μάλλον θα πρέπει να μιλάω λίγο πιο σιγά. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε ότι έχουμε και πάλι τους ίδιους ε, ακτιβιστές που διαδίδουν τις πληροφορίες αυτές. Θα πρέπει λοιπόν να το κατανοήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Από τη Γερμανία, για παράδειγμα, βλέπετε και πάλι τη Συρία. Δύο γαλλικές εταιρείε στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε την FADH που είναι υπεύθυνη για την FIDH σε ό,τι αφορά ε, αποφάσεις για το κατά πόσο είναι το νόμιμη ή όχι χρήση κάποιων προϊόντων. Πώς έχουμε φτάσει λοιπόν εδώ και πώς έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση που χρειάζεται να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Στην επόμενη διαφάνεια κατήσατε σαφές ότι ε, σε όλα αυτά τα μέρη του κόσμου εξαγάγεται ε, ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκά προϊόντα παρακολουθήσεις και βλέποντας λοιπόν ε, πώς συμβαίνουν αυτά βλέπετε μία επισκόπηση εδώ στη διαφάνεια αυτή για το πώς είναι οι ρυθμισμένοι εξαγωγές προϊόντων παρακολούθησης και μη ρυθμισμένες εξαγωγές. Βλέπετε λοιπόν το τι με κόκκινο χρώμα τις ε, εγκεκριμένες, τις ε, εξαγωγές με άδειε. Συγγνώμη, τα κόκκινα προϊόντα είναι μία μόνο ε, εταιρεία που εξαγάγει λοιπόν προϊόντα η οποία πιστεύω ότι δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία και έχουν διαρρεύσει αυτά στο διαδίκτυο πλέον. Με το μπλε χρώμα βλέπετε τις ελεγχόμενες και αδεδεδεμένες εξαγωγές. Στην επόμενη διαφάνεια λοιπόν βλέπετε ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο φαινόμενο. Αυτό αφορά όλες τις χώρες. Βλέπετε λοιπόν την, ε, την ισιακή υποδομή παρακολούθησης ε, και φαίνεται με σαφήνεια ότι οι ευρωπαϊκές εταιρείες ε, μπλέκονται σε κάθε επίπεδο. Βλέπετε λοιπόν υπάρχουν διάφορα επίπεδα από το web filtering μέχρι και τις επιθέσεις hacking και σε όλες τις φάσεις η Τινησιακή Κυβέρνηση έλαβε υποστήριξη από ευρωπαϊκές εταιρείες και από διάφορους φορείς όχι μόνο για να εξαγάγει, αλλά για να υποστορίξει και να, να συντηρήσει τα συστήματα αυτά. Είναι λοιπόν λυπηρό που στις περιπτώσεις αυτές ε, ακόμα και έκπτωση είχαν για να μπορούν να ε, ελέγχουν και να δοκιμάζουν τα συστήματα στο ευνησιακό σύστημα. Αυτή ήταν λοιπόν η κατάσταση μέχρι πριν από κάποιες εβδομάδες, μέχρι να κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγέ. Τι τελευταίες τρει λοιπόν εβδομάδες υπάρχει ένα διαφορετικό πλαίσιο για τον έλεγχο των ε, εξαγωγών. Άρα, γιατί να μας απασχολεί αυτό, γιατί να σας απασχολεί εσά τα μέλη των επιτροπών σας. Νομίζω ότι είναι σαφές ε, και χάρη στην κυρία Σχάκη και την κυρία Λοχμπίλερ που προωθούν το θέμα αυτό και έχουν ηγετικό ρόλο στην επιτροπή αυτή. Αν όλα είναι, παρακολουθούνται, τι διαφορά έχει η επιπλέον ε, τεχνολογία. Νομίζω ότι πλέον αυτό που διαφέρει είναι ότι έχουν ε, αρχίσει να μιλούν τα θύματα και λένε, μας δείχνουν τι έχει συμβεί και ότι έχουν φωνή και στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε έχουμε και καλύτερη τεκμηρίωση που καταδεικνύει ποιο είναι ο αρνητικό αντίκτυπο τη ε, παρακολούθηση. Και έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε σιγά σιγά τι τεχνολογίε τη Ευρώπη, τι αντίκτυπο έχουν ε, στι τρίτε χώρε και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Και θα πρέπει να προσθέσουμε ότι υπάρχει μια συμμαχία διάφορων ΜΚΟ που φαντάζομαι ότι βρίσκονται και εδώ στην αίθουσα και θα μιλήσουν στο δεύτερο τμήμα του πάνελ για που ασχολούνται με τα θέματα αυτά και που αρχίζουν να κατανοούν ε, τον αντικτύπο και τις ε, βλάβες που προκαλούνται. Και αυτό έχει αλλάξει σημαντικά και την πολιτική. Στα τέλη του 2013 η ρύθμιση του Βάσεναρ προσπάθησε να συμπεριλάβει στις λίστες της, στους καταλόγους της και τα θέματα προϊόντων παρακολούθησης. Έγινε μια συζήτηση για τους ορισμούς. Είναι μια απόπειρα να ανταποκριθούμε σε αυτές τις προκλήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώνει το σχετικό κανονισμό για τα προϊόντα της χρήσης και κάνει μια σημαντική συζήτηση και με τη βιομηχανία. Αυτή η συζήτηση έχει γίνει μία από τις συζητήσεις κλειδί για την μεταρρύθμιση της σχετικής νομοθεσίας και νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει το πόσο σοβαρή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και στο εμπόριο αλλά και στις εξωτερικές σχέσεις. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ε, εταιρείε που το κάνουν αυτό. Αλλά τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει καταδεικνύουν ότι ακόμα και οι πιο, μεγάλες, ε, πιο μεγάλοι παραβάτες, αν θέλετε, της νομοθεσίας αυτής προσπαθούν με κάποιο τρόπο να ανταποκριθούν στις νέες συμβατικές σχέσεις με τρίτες χώρες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αλλάζουν σιγά σιγά τα πράγματα. Υπάρχει μία απόπειρα να αλλάξουν. Φυσικά η κατάσταση δεν είναι ιδανική, δεν είναι φανταστική, δεν πρόκειται να υποστηρίξω κάτι τέτοιο και νομίζω ότι το πιο σημαντικό ζήτημα είναι η διαφάνεια. Όλες οι συζητήσεις για τις εξαγωγές γίνονται κυκλισμένων των θύρων ε, ουσιαστικά. Αυτό δεν γίνεται απαραίτητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, γιατί επιμένουμε, αλλά σίγουρα αυτό γίνεται στα πλαίσια του Βασενάρ. Και τελικά δεν ξέρουμε τελικά, ποτέ ποιο είναι υπεύθυνο. Χρειάζεται λοιπόν λογοδεσία και διαφάνεια. Γίνονται φυσικά διεθνεί διαπραγματεύσει, αλλά κάπω θα πρέπει να εμπλακεί και η κοινωνία των πολιτών στην όλη διαδικασία για να κατανοούν και οι πολίτε τι γίνεται. Πέρα από αυτό, στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε το όλο θέμα τη κρυπτογράφηση. Νομίζω ότι δεν θα επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Είναι σημαντικό ωστόσο να υπογραμμίσουμε ότι οι έλεγχοι προϊόντων της χρήσης προσπαθούν να ελέγξουν την κρυπτογράφηση. Θεωρώ ότι αυτό είναι παράλογη, παράλογος περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όταν ε, καταλάβουμε ότι η κρυπτογράφηση είναι ένας από τους λίγους τρόπους που έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του για να προστατευτεί από τη μαζική παρακολούθηση. Η κρυπτογράφηση λοιπόν είναι ο μοναδικός τρόπος που έχει ένα άτομο να προστατευτεί είναι λοιπόν παράλογο να προσπαθούν οι κυβερνήσει να το ρυθμίσουν αυτό. Ένα τελευταίο ε, σημείο πέρα από τους ορισμούς ε, στην επόμενη διαφάνεια. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ορισμοί που κυκλοφορούν και συζητιούνται στα διάφορα φόρα. Η Βάσιναρ μιλάει για cyber tools, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για τεχνολογίες ε, ανθρώπινης ασφάλειας, Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι ορισμοί που καλύπτουν διαφορετικέ έννοιε και όταν γίνονται οι συζητήσει, για το τι ρυθμίζουμε θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε όσο πιο σαφεί γίνεται. Ποιο θέλει να ρυθμίσει τι και πώ είναι και σαφεί και αποτελεσματικοί οι ορισμοί προκειμένου να προστατεύουν όντω τα ανθρώπινα δικαιώματα στα πλαίσια τη γενικότερη εμπορική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, όπω είπε και ο πρόεδρο, δεν θα πρέπει να επιτρέπει να γίνονται παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω εξαγωγή προϊόντων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Σα ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Πάρα πολύ γρήγορη και εξαρτητική παρουσίαση. Και τώρα να δώσω το λόγο στον Κρίστιαν Χόιχερτ, ο οποίος είναι σύμβουλος IT και μέλος του Cars Computer Club στη Γερμανία. Um, I have written speech, so um, I read that from paper. the <coughs> members of European Parliament, Ευχαριστώ, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκλησή σας. Από το 1981 τίθεται θέμα ελευθεριών του πολίτη και χαιρόμαστε που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό των ψηφιακών τεχνολογιών και των ελευθεριών του πολίτη. Εγώ θα σας μιλήσω για τα Πρόβλημα με το εύρος, πρόβλημα με τη, τους ορισμούς, με τον έλεγχο των εξαγωγών και σίγουρα υπάρχουν λόγοι για ανησυχία σήμερα αρκετοί. Το θέμα του εύρους. Πρέπει να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Είναι περίπλοκο όταν μιλάμε για τη μεταφορά τεχνολογιών που έχει να κάνει με την ασφάλεια στο σημερινό κόσμο. Επειδή βασίζεται στις συζητήσεις μας, πολύ συχνά βλέπουμε ότι είναι ένα πρόβλημα που δεν το καταλαβαίνουμε καλά όταν συζητάμε. Η έρευνα έχει να κάνει με την αντοχή των διαφόρων συστημάτων πληροφορικής προκειμένου να μειωθεί η ζημιά που μπορεί να προκαλέσουν. Στην έρευνα λοιπόν πρέπει να έχουμε πραγματικά παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Η παρεμβολή επίση παίζει ένα σημαντικό ρόλο στις, ε, στην έρευνα. Η χρήση των ε, μέσων που χρησιμοποιούμε εξαρτάται από το τι προβλήματα θέλουμε να αναλύσουμε. Πολύ συχνά θέλουμε να δείξουμε στους πελάτες τι πρόβλημα μπορεί να προκληθεί από τις δράσεις τους. Δεν φτάνει να τους λέμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Για να λυθούν τα προβλήματα πρέπει να υπάρχει ένας κώδικας πριν γίνει η διανομή. Κάτι το οποίο βέβαια κοστίζει και σε χρήμα και σε χρόνο. Αλλιώς ο χρήστης, ο πελάτης, δεν θα αντιδράσει με το σωστό τρόπο. Ένας από τους πιο βασικούς τρόπους για να λύσουμε τα σημερινά προβλήματα είναι να έχουμε ισχυρά software. Αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να μπορούμε να τα σπάσουμε, να μπούμε μέσα δηλαδή. Πώς λειτουργεί πραγματικά η ασφάλεια. Και έτσι φτάνουμε στη δεύτερη ανησυχία που είναι το θέμα των ορισμών Η σημερινή ενημέρωση όσον αφορά τους ελέγχους μας φέρνει κοντά σε διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούνται, μηχανικής και άλλες. Το software προσπαθεί να βρει για παράδειγμα πόσο αποτελεσματική είναι η παρεμβολή. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται από εκείνους οι οποίοι μπορούν να χειριστούν τα διάφορα λειτουργικά συστήματα. Και μη κυβερνητικέ οργανώσεις και κυβερνήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η παρεμβολή μπορεί να είναι αποτελεσματική και να δείξει πού υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας. Ένας καλός ορισμός μπορεί να έχει να κάνει με την δυνατότητα να εντοπίσουμε στόχους. Η παρακολούθηση σημαίνει ότι έχουμε δεδομένα τα οποία δεν μπορούμε να τα αναλύσουμε απαραίτητα. Πρόκειται για μια ιδιοκτησία δηλαδή που χρησιμοποιούμε χωρίς να έχουμε την άδεια. Δεν καθορίζεται όμως πάντα επαρκώς. Οπότε καταχρώμαστε κατά κάποιο τρόπο την ιδιοκτησία του άλλου με την παρακολούθηση. Οι έλεγχοι εξαγωγών ορίζουν την τεχνολογία για το software παρεμβολής και πώς πρέπει να ελέγχεται. Η εισβολή μπορεί να βοηθήσει προκειμένου να αναπτύξουμε περισσότερο την ασφάλεια. Ο έλεγχος των τεχνολογιών πάντως, ανάπτυξη software, είναι κάτι πολύ ευρύ και αντιτίθεται στις αρχές της ίδιας μηχανικής αυτής καθ' αυτής. Χρειάζεται βελτίωση της ασφάλειας που έχει όμως νόημα. Η έρευνα για την ασφάλεια πλήττει τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε τρίτες χώρες. Αυτό σημαίνει ότι τελικά παγκοσμίω τίθεται το θέμα αυτό της έλλειψης ασφάλειας. Ό,τι κάνουμε εδώ επηρεάζει και το τι γίνεται σε τρίτες χώρες. Και έτσι ερχόμαστε στο τρίτο κομμάτι που λέει τι μαθήματα έχουμε πάρει από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Για να καταλάβουμε πώς οι έλεγχοι των εξαγωγών επηρεάζουν την ασφάλεια στην τεχνολογία, πρέπει να δούμε τι έγινε με τα crypto που είχαμε τη δεκαετία του 90 με την αποκρυπτογράφηση των επικοινωνιών. Ο έλεγχος των εξαγωγών και η αποκρυπτογράφηση επηρέασε πολύ την κατάσταση την εποχή εκείνη και τα αναπτύχθηκαν πολύ περισσότερο τα πρωτόκολλα, διάφορες συμφωνίες. Πώς Τώρα την εξαγόμενη αποκρυπτογράφηση την χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιείται καινοτομία στον τομέα των επικοινωνιών και οι έλεγχοι των εξαγωγών σίγουρα θα έχουν περισσότερο αρνητικές συνέπειες στην ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής στο μέλλον και εδώ και αλλού. Εν κατακλείδη. Προκειμένου το software να είναι ασφαλές, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα παραδείγματα και εργαλεία. δεν πρόκειται για δύο του ίδιου νομίσματος, το πώς δηλαδή θα ασφαλίσουμε ένα software ή πώς θα το σπάσουμε. Θα έλεγα ότι πρόκειται για το ίδιο νόμισμα, απλώ για την ίδια όψη του νομίσματος. Αν πιστεύετε ότι οι έλεγχοι εξαγωγών κάνουν περισσότερο καλό παρά κακό, προτείνουμε να γίνεται διάκριση της παρεμβολής από την ε, κατάχρηση. Χρειάζονται... Χρειάζεται τέλος να έχουμε υπόψη μας την ελευθερία του λόγου. Αν μιλάμε για κώδικα, και περί αυτού πρόκειται ουσιαστικά, δεν πρόκειται μόνο για τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, πρόκειται για την ελευθερία του λόγου. Ένα, κακό, ένα συγγνώμη, θετικό, ένα καλό, το οποίο δεν μπορούμε να εμπορευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Χάιχαρτ. Είδαμε λοιπόν και την πλευρά του χρήστη, είδαμε και την πλευρά των επιστημόνων για την ελεύθερη χρήση του λογισμικού και τώρα θα ακούσουμε και την πλευρά της βιομηχανίας ε, και καλωσορίζω τον κύριο Μάγνους Νόρντεϊς ε, ο οποίος ε, είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο εξαγωγών της Digital Europe. Ευχαριστώ πολύ αγαπητή συμπρόεδρε, η κυρία Βαλενσιάνο, κυρία, κύριε Λάγκε. Ε, ε, ε, συμμετέχοντες μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πολυπληθές το ακροατήριο εδώ λέγομαι Μάγνους Νορντέους και εδώ εκπροσωπώ την βιομηχανία της ψυχιφιακής τεχνολογίας στην Ευρώπη όπως είπε και ο κύριος Λάγκε είμαι issue manager για τις του ελέγχους των εξαγωγών της Digital Europe και επίσης ε, είμαι και ε, νομικός σύμβουλος για την εμπορική πολιτική και τη συμμόρφωση ε, της Σουηδικής εταιρείας Ericsson η ε, ε, τεχνολογία της πληροφορίας, τεχνολογία της επικοινωνίας ε, και οι τομείς ε, των ε, ηλεκτρονικών αγαθών, καταναλωτικών αγαθών είναι θέματα τα οποία απασχολούν την Digital Europe. Εμείς εκπροσωπούμε 59 διεθνείς εταιρείες, 36 διεθνείς εμπορικές ενώσεις και περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις με 2 εκατομμύρια υπαλλήλους. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ε, ε, ε, πω δύο λόγια όσον αφορά την αναθεώρηση της πολιτικής ελέγχου των εξαγωγών. Βλέποντας την σημερινή κατάσταση όσων των κρατών μελών και τον τραχή ανταγωνισμό όσον αφορά την σφαιρική βιομηχανία είναι σημαντικό ε, να ε, γίνουν έλεγχοι εξαγωγών ε, όσον αφορά τα πιο ευαίσθητα προϊόντα ενώ τα λιγότερο ευαίσθητα θα μπορούν να έχουν ελεύθερες εξαγωγές ή πιο ελεύθερες εξαγωγές. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της λεγόμενης γενικής αδειοδότησης εξαγωγών ε, και βεβαίως η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματο αυτού μπορεί να παίξει πάρα πολύ σημαντικό ε, ρόλο. Κατά την άνοια αυτή εμείς ε, ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη της μια ευρύτερη σειρά αδειοδοτήσεων γενικών εξαγωγών ε, κυρίως όσον αφορά την κρυπτογράφηση, τους ε, ημιαγωγούς, καθώς επίσης ε, και τις μεταφορές εντός των ομίλων και εντός των εταιριών, ας πούμε, μέσα από την έρευνα και ανάπτυξη. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο, ρόλο προτύπου, μοντέλου, όσον αφορά τον, το σύστημα ελέγχου συνολικών σφαιρικών εξαγωγών και να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή η βιομηχανία μπορεί ε, να ε, δώσει μεγάλη όθηση στον τομέα μέσα από τα εσωτερικά της ε, προγράμματα συγγνώμη, συμμόρφωσης το σύστημα ελέγχου των εξαγωγών μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά και αποτελεσματικά στην διεθνή αγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, για την ε, δέσμευση, την στράτευση την οποία έχετε όσον αφορά αυτό το εξαιρετικά ε, σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε τους ελέγχους των εμπορικών συναλλαγών καθώς επίσης και το ενδεχόμενο ακόμα και οικονομικών κυρώσεων από αυτή την άποψη. Πέρα από την παραδοσιακή φύση του ελέγχου των εξαγωγών εκλογών ε, ε, ως ε, μέσο αποφυγής της χρήσης τεχνολογιών για κακό σκοπό πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και, και τελευταίες εξελίξεις όπως ας πούμε τα Wikileaks και τα λοιπά. Ε, πιστεύω ότι ε, μάλλον θα πρέπει να σημειώσω ότι η Digital Europe ε, είναι απολύτως δεσμευμένη όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει και δικά της εσωτερικά συστήματα τέτοιου ελέγχου. Ωστόσο, είμαστε πεπισμένοι ότι η μεγαλύτερη συμβολή ε, μπορεί να γίνει μέσα από την ίδια την ψηφιακή τεχνολογία ε, και επίσης πιστεύουμε ότι οι επικοινωνίες και η συνδεσιμότητα ε, μπορεί να δώσει απάντηση σε βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε το 2012 ε, στο Digital Freedom Statement ε, ε, οι τεχνολογίες πληροφόρησης και πληροφορίες και επικοινωνίας έχουν υπάρξει σημαντικές στην οργάνωση κοινωνικών κινημάτων και εξεγέρσεων σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να δούμε και να αναλύσουμε ακόμα πιο προσεκτικά ε, αυτές ε, τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας για τις οποίες θα πρέπει να δημιουργήσουμε νέα στάνταρ και νέες δυνατότητες ελέγχου έστω και αν αυτό είναι αρκετά δύσκολο όπως ανέφεραν οι προλαλήσαντες. Όταν μιλάμε για νέους ελέγχους, κυρίως όταν αυτοί είναι μονομερείς, είναι απόλυτης σημασίας ε, αυτοί οι νέοι έλεγχοι να έχουν ε, οργανωθεί με σωστό τρόπο έτσι ώστε ο αντίκτυπος των ελέγχων αυτών να είναι απολύτως ε, σαφής έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε από μόνοι μας εμπόδια στις στο εμπόριο που τελικά δεν θα, θα έχουν μόνο υψηλό κόστος για όλους και κανέναν σημαντικό αντίκτυπο. Ε, μερικές φορές ε, φαίνεται εύκολο να λυθούν ε, κάποια προβλήματα μέσα από τον έλεγχο των εξαγωγών. Εγώ λέω ότι θα πρέπει απλώς να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακριβώς για την ψηφιακή παρακολούθηση και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να εξάγουμε αυτά τα συστήματα τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν ένα καλό σύστημα τηλεπικοινωνιών χωρίς να αφήνουν δίνουν μεγάλες δυνατότητες σε ε, πρακτικές ε, ε, παρίσδησης ή παρακολούθησης. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν είναι σημαντικό να δούμε και εναλλακτικέ λύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν πολύ πιο σφαιρική κάλυψη χωρίς να εγείρουν αντιφάσεις και αντιφατικές, αντιφατικούς αντικτύπους. Ε, πιστεύουμε ότι η γεωγραφική κάλυψη, ας πούμε, είναι ε, πάρα πολύ σημαντική. Όταν ε, μιλάμε για νέους ελέγχους ελπίζουμε ότι το μήνυμα θα είναι σαφές. Η ψηφιακή τεχνολογία και η βιομηχανία της στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν πάρα πολύ σκληρό ανταγωνισμό από ανταγωνιστές από τρίτες ε, χώρες και επομένως οποιασδήποτε νέες μορομερείς προσπάθειες ελέγχου των εξαγωγών από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργήσει ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα. Ε, είναι γεγονός ότι οι διευρυμένοι έλεγχοι των εξαγωγών μπορούν, μπορεί να έχουν υψηλό κόστος για την ευρωπαϊκή βιομηχανία ε, και στο τέλος ε, να έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στις θέσεις απασχόλησης αλλά και στην ανάπτυξη. Εμείς βεβαίως θέλουμε να υπάρχει έλεγχος αλλά θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει προσεκτικά σε αυτή τη φάση της προπαρασκευής του νέου κανονισμού όλες τις πλευρές και την πλευρά των, και του κόστους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Βεβαίως, εμείς στηρίζουμε την αναθεώρηση ε, της ε, ε, πολιτικής των εξαγωγών και λέμε ότι πραγματικά όσον αφορά την αποκρυπτογράφηση, του ημιαγωγούς και τις εμβετερικές μεταφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ειδική μέρημνα. Θα παρακολουθούμε από κοντά και θα είμαστε και εμείς αρρωγοί στη διαδικασία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και τώρα έχουμε ε, προβλέψει συζήτηση με τους βουλευτές. Δεν έχω κανέναν όμως που να έχει ζητήσει το λόγο. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Με προκαλεί έκπληξη. Ο κύριος Ρούμπιχ όμως ζητάει το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές παρουσιάσεις. Θα ήθελα να υποδείξω ότι και στο Κοινοβούλιο Στην αξιολόγηση των ε, επιστημονικών δυνατοτήτων έχουμε κάνει σχετική μελέτη για τη μαζική παρακολούθηση που ασχολείται με τα τεχνικά ζητήματα και θα σας σύστηνα να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μελέτη γιατί εκεί υπάρχουν σαφείς ορισμοί για τους διάφορους τομείς και νομίζω ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για την εργασία σας στο μέλλον, για την πρακτική εργασία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Λίγο Η επόμενη ομιλήτρια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλους τους πανελίστες που ήρθαν εδώ στις επιτροπές μας και κατέβαλαν τον κόπο να κάνουν τις παρουσιάσεις. Καταρχάς, μία παράκληση θα ήταν δυνατόν να λάβουμε τις ε, παρουσιάσεις σας γιατί δεν χρειάζεται άλλωστε να μας ε, δώσετε σε όλες τις γλώσσες, μόνο τα αγγλικά. Μια δεύτερη ερώτηση, η οποία προέρχεται από την έλλειψη γνώσεως, γιατί δεν είμαι ειδική καθόλου ε, στα θέματα αυτά. Αλλά έχω παρόλα αυτά την αίσθηση ότι όλες αυτές οι τεχνικές, όλη αυτή οι στόχοι, να, η πρόθεση να ελεγχθεί ένα συγκεκριμένο κλάδος όσο και αν είναι σωστή έχει αντικτυπώ και σε άλλους τομείς για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Δεν βλέπω λοιπόν απόλυτα πώς αυτό μπορούμε να το διαχωρίσουμε επακριβώς. Αν δεν θέλει κάποιο θεσμικό όργανο να το διαχωρίσει. Ίσως θα μπορούσατε να με καθησυχάσετε, να με εξηγήσετε, εν πάση περιπτώσει. Trying to Η κυρία Σχάκη. Ε, Προσπαθώ να ακούσω, προσπαθώντας να ακούσω τους δύο συναδέλφους. Opposite things. Ένα... νομίζω ότι λένε αντίθετα πράγματα και εδώ κάτι θα πρέπει να με εξηγήσετε παραπάνω, γιατί ε, εγώ καταλαβαίνω ότι ασχολούμαστε με τα προϊόντα της χρήσης, ότι εξαγάγουμε τέτοια λογισμικό παρακολούθηση στην Αίγυπτο, την Τινησία, σε χώρες όπου υπάρχει καταπίεση των ακτιβιστών ή υπήρχε τουλάχιστον στο παρελθόν ε, και θεωρούσαμε ότι κάναμε κάτι το σωστό. Και άκουσα και τον κύριο Μπόρχερ, το οποίο μα είπε ότι αυτό ουσιαστικά δεν είναι καλό. Δεν είναι καλή ιδέα. Για να προσπαθήσουν λοιπόν αυτές, αυτοί οι δύο πανελίστες να μας εξηγήσουν σε μια γλώσσα κατανοητή, χωρίς bits και bytes, σας παρακαλώ γιατί είναι ένα βασικό θέμα αυτό και ειλικρινά δεν το κατάλαβα. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, κυρία Ροντρίγκες. Ευχαριστώ πολύ για τις ε, παρουσιάσεις σας. Και εγώ είχα λίγο αυτή την ίδια αίσθηση με την συνάδελφο γιατί έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα τμήμα αυτόν που ακούσαμε που ε, ε, έρχεται σε αντίθεση με αυτά που ακούσαμε ε, από, τους, από τον άλλο μιλητή όσον αφορά την χρήση των τεχνολογιών και την εξαγωγή τους. Θα ήθελα λοιπόν λίγο να εμβαθύνουμε γιατί φυσικά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποιο θετικό δυναμικό το οποίο μπορεί και πρέπει να προωθηθεί αλλά χωρίς να λησμονούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα γιατί αυτό μας ενδιαφέρει εδώ.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 θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες συνάδελφοι. Νομίζω ότι υπάρχουν στοιχεία αντίφασης ε, στις πληροφορίες και τις παρεμβάσεις που ακούσαμε. Εγώ πιστεύω ότι η εστίαση της συζήτησης, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, ε, θα πρέπει ε, να είναι οι ενδεχόμενες αντιφάσεις που μπορούν να υπάρχουν από, ανάμεσα αφενός τις εμπορικές συμφωνίες και αφετέρου στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να εστιάσουμε τις ε, ε, συζητήσεις μας ε, και να συζητήσουμε και συγκεκριμένα για συμφωνίες τις οποίες συζητούμε τώρα, αυτή τη χρονική περίοδο. Θα ήθελα ας πούμε να καταλάβω στα πλαίσια της συμφωνίας TTIP με τις Ηνωμένε Πολιτείε. τι θέση έχει αυτή η συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνάδελφος Αστραβίτσιος. Thank you. ευχαριστώ. Καλημέρα και ευχαριστώ και εγώ για τις παρουσιάσεις σας. Εξαιρετική, εξαιρετική εισαγωγή στον νέο κόσμο που τεχνολογίες που μας βοηθούν να επιζήσουμε σε αυτό τον περίπλοκο κόσμο. Από την άλλη μεριά όμως μας φέρνουν μπροστά σε νέους κινδύνους και νέες προκλήσεις σε τι βαθμό η συνεργασία των ευρωπαϊκών ε, επιχειρήσεων που συνεργάζονται μεταξύ τους, ε, συνεργάζονται και με τον τρίτο κόσμο, ε, επιχειρήσεις οι οποίες αναπτύσσονται πολύ γρήγορα και έχουν όλο, συλλαμβάνουν όλο και περισσότερες ιδέες, καινοτόμε ιδέες σε αυτό το τομέα. Τι κίνδυνο βλέπετε εσείς από τη συνεργασία αυτή. Όχι απαραίτητα επίσημη συνεργασία με επιχειρήσεις από τρίτες χώρες, Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα. Ο κύριος Πάλο Βρατσότη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους αξιότιμους ευρωβουλευτές και το πάνελ. Πρώτα απ' όλα, από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέλουμε να επικεντρωθούμε περισσότερο στα κοινά που έχουμε με αυτούς που πήραν το λόγο. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες, το θέμα της παρακολούθησης, της παρίσδησης και της σχέσης τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να επικεντρωθώ στα όσα έχουμε ήδη κάνει. Ο κύριος Βάγκνερ αναφέρθηκε σε αυτό. Πράγματι εδώ και μερικές εβδομάδες έχουμε προχωρήσει με έναν κανονισμό και φαντάζομαι ότι θα καταφέρουμε να μακρύνουμε και την πλεγραμμή που δείξατε στο διάγραμμα και να την φτάσουμε στην κόκκινη. Αυτό που είπαν όλοι, ότι αλλάζουν οι έλεγχοι, δεν γίνονται όπως γινόντουσαν κάποτε, τώρα γίνονται έτσι ώστε η τεχνολογία high-tech δεν θα περάσει από τους καλούς τους κακούς. Τώρα είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Χρειαζόμαστε πιο ευέλικτη προσέγγιση. Και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την ε, κυρία Σχάκε για τα πολύ σημαντικά που είπε για την αναθεώρηση του κανονισμού. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Έχουμε αναθεώρηση του κανονισμού ε, για τη ρύθμιση των εξαγωγών Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή και με την επιστημονική κοινότητα για να βασίσουμε σε επιστημονικά δεδομένα τον κανονισμό μας και να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται καλύτερη γνώση. Για την ε, ελαστικότητα τώρα και την ευελιξία, όπως είπατε, αν προσπαθείτε να τα βρείτε όλα και να τα παρακολουθήσετε όλα, τότε θα γεμίσετε από πράγματα τα οποία μπορεί να είναι και άχρηστα. Οι Αμερικανοί είναι καλοί τα και έχουν και ένα άλλο που λέει ότι πρέπει να χτίζουμε ψηλούς φράχτες γύρω από ένα μικρό κήπο. Αυτό έχει να κάνει με τις γενικές αδειοδοτήσεις και με την προσπάθεια να μην μπούμε σε παράνομο εμπόριο. Η αντίφαση στην οποία αναφερθήκατε έχει να κάνει κυρίως με το ότι είναι πολύ δύσκολο να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε να ελέγξουμε. Εδώ είναι που χρειάζεται η πραγματογνωμοσύνη. Εμείς έχουμε ειδικού και συνεργαζόμαστε και με τους ειδικού από τις χώρες μέλη, με τον κλάδο. Προσπαθούμε να βασιστούμε στην εμπειρία που έχουμε μέχρι τώρα για να κάνουμε καλή δουλειά οι ενδιαφερόμενες πλευρές, οι έμποροι, οι κυβερνητικέ οργανώσεις, όλοι αυτοί μπορούν να μας ενημερώνουν και φροντίζουμε να μας ενημερώνουν και να μας πληροφορούν ώστε να είμαστε και εμείς σε θέση να αντιμετωπίζουμε τις απειλές. Για τον έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αν δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι άλλοι θα το κάνουν. Είναι όλο και περισσότερο προφωνές ότι για να συμμετέχουμε παγκοσμίως στον κλάδο της ε, τεχνολογίας εχμής ε, πρέπει να συμμετέχουμε. Δείτε τι κάνει η Κίνα. Προσπαθούν ακόμα και αν ε, δεν συμμετέχουν στο σύστημα κάνουν και αυτοί πράγματα. Και ένα άλλο σχόλιο για το TTIP και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει και αυτό παρόλο που δεν είναι αντικείμενο αυτής της συζήτησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την ευκαιρία αυτή, για αυτή την ακρόαση και προσβλέπω σε συνεργασία με όλους σας στο μέλλον. σε ευχαριστούμε. Τρία λεπτά τώρα για να απαντήσουν ο κύριος Βάγνερ πρώτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για να απαντήσω στα διάφορα σημεία που αναφέρθηκαν. Νομίζω ότι αυτά που συζητήσαμε εδώ ε, προκαλούν και έχω μεγαλύτερη ελευθερία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσω για τέτοια θέματα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε ό,τι αφορά το εμπόριο, ε, ότι θα υπάρχει γενική αποδοχή για το πώς λειτουργεί το, εμπόριο και πώς ε, δράει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο διεθνές προσκήνιο και νομίζω ότι ήταν σωστό και αυτό που ανέφερε και κάποιος άλλος βουλευτής. τα ανθρώπινα δικαιώματα ενδεχομένω υπάρχει κίνδυνο να θεωρηθούν ε, υποκείμενα στα εμπορικά συμφέροντα. Τα ανθρώπινα δικαιώματα όταν εφαρμόζονται σωστά στην, ε, ε, στο εμπόριο αυξάνουν την νομιμότητα του εμπορίου, δεν το εμποδίζουν. Και νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να βρούμε μια σημαντική ισορροπία, αυτά που είπε η κυρία Σαρτζεντίνη για την ε, βασική διαφωνία μεταξύ των εισηγητών. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλη η διαφωνία όσο φαίνεται. Εμείς ε, κοιτάμε θέματα κρυπτογράφησης και επίσης βλέπουμε και θέματα που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ύστερα πτύχονται και θέματα ε, τεχνολογικά. Ποια τεχνολογία θα πρέπει να χρησιμοποιείται και ποια όχι. Και συμφωνώ με αυτά που λένε κάποιοι ερευνητέ ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ακόμα πνευτότητα έρευνα και ανάπτυξη. Το πώ θα εφαρμόζεται αυτό από εμά και από τα κάτι μέλη είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να επιλέξω, αλλά νομίζω ότι ακούγοντα αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά συμβαίνουν, αυτό γίνεται. Αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η εφαρμογή του κανονισμού που ισχύει εδώ και τρία, τρεις εβδομάδες θα συνεχιστεί σωστά. Να μην ξεχνάμε όμως και πώς θα βελτιώσουμε την αποδοχή του διεθνούς εμπορίου. Εξασφαλίζοντας ότι θα γίνουν αποδεκτές ρυθμίσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να μην βασιστούμε αποκλειστικά στην άποψη της βιομηχανίας ή να μην επικεντρωθούμε υπερβολικά στο πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι σε όλες τις καταστάσεις αυτό που ε, κάνουμε θα θεωρηθεί αποδεκτό. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής. Υπάρχουν κάποιες διαφορές ε, άποψης γιατί εμείς πιστεύουμε ότι η ουσία έγκυται στον ορισμό. Ο διαχωρισμός ασφαλούς και μη ασφαλούς λογισμικού είναι ε, πάρα πολύ δύσκολος Ε, κάθε μηχάνημα μπορεί να έχει ε, πάρα πολλές δυνατότητες λογισμικού και επομένως ε, υπάρχουν και πολλές δυνατότητες ελέγχου. Από την άλλη πλευρά η ε, ε, παρεμβολή ή η η παρισδηση intrusion είναι ένα στοιχείο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αλλά είναι και μια δυνατότητα προστασίας του λογισμικού. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πάρα πολλοί νόμοι σε όλες τις χώρες. Στη Γερμανία είναι εξαιρετικά πολλοί και λεπτομερείς οι νόμοι οποίοι αφορούν αυτήν την ασφάλεια και προς είναι. η ανασφάλεια ή η ανασφάλεια του λογισμικού ε, και των υπολογιστών είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα τα οποία έχουμε ε, τα θέματα τα οποία σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στην ουσία αυτά τα ίδια ζητήματα τα οποία αφορούν ε, την γενικότερη ασφάλεια του, του λογισμικού. Όταν μιλάμε για intrusion software ε, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να δούμε κάποιες άλλες παραμέτρους οι οποίες μας οδηγούν σε κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες όμως δεν αρκούν έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Η λύση φυσικά δεν είναι να σταματήσουμε ε, να εμπορευόμαστε ε, αυτά τα ε, εργαλεία γιατί δεν ασχολείται μόνο η βιομηχανία με αυτά, ασχολείται και το πανεπιστήμιο, ασχολούνται και τα παιδιά τα οποία παίζουν με τους υπολογιστές συνέχεια. Και επομένως νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιες είναι και οι επιπτώσεις ε, ε, αυτών των διαδικασιών. Στην Γερμανία είχαμε ας πούμε ε, το WG και όπου κόπηκαν όλες οι εξαγωγές οι οποίες δεν συμμορφώνονταν με τους κανονισμούς του ελέγχου των εξαγωγών. Ε, ε, ε, και, και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μας λένε δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς σε ποιο κανονισμό δεν συμμορφωνόμαστε και δεν καταλαβαίνουμε ακριβώς που έγκυται η μη συμμόρφωση και υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες ε, έχουν σαν κύριο στόχο ε, την ε, επίθεση εναντίον συστημάτων ή ανθρώπων και που βρίσκουν την δυνατότητα να ξεπεράσουν τα προβλήματα ακριβώς λόγω της ασάφειας που υπάρχει. Ο έλεγχος των εξαγωγών που έχει γίνει μέχρι τώρα δεν έχει οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να αλλάξει λοιπόν, να πάμε στο αντίθετο άκρο. Ο κύριος Μάγνους Νόρντεους, ε, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι πάρα πολύ περίπλοκο το να ε, νομοθετήσει κανείς για το θέμα αυτό. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε, όπως όλοι συμφωνούμε ε, επί της σημασίας που έχει η σωστή νομοθέτηση. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά συμβάλαμε ε, σε μία μελέτη του Ινστιτούτου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επιχειρηματικότητα ε, με το θέμα αυτό δεν είναι δυνατόν ας πούμε να ε, επιβάλλει κανείς περιορισμούς ε, στο, στο διαδίκτυο και τη χρήση διαδικτύου σε μία άλλη χώρα. Ε, είναι πολύ σημαντικό επίσης οποιαδήποτε μέτρα και αν πάρει κανείς να μην παρεμβάλλεται στην ασφάλεια και την πληρότητα του συστήματος τηλεπικοινωνιών μιας άλλης χώρας. Εμείς στα Telecom έχουμε μία σειρά θεμάτων τα οποία είναι υποχρεωτικά για κάθε ε, δίκτυο και πιστεύουμε ότι ε, αυτά θα πρέπει ε, να μπορούν να παρέχονται από τη μία αγορά στην άλλη οι εταιρείε Ευρωπαϊκής, που έχουν βάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βεβαίως ε, έχουν την υποχρέωση και το κάνουν να ενσωματώσουν δηλαδή ε, το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις, στα συστήματα τα οποία αναπτύσσουν και εμπορεύονται είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει ένα και μόνο σύστημα συνολικού ελέγχου των εξαγωγών. Έχουμε 1,2 εκατομμύρια ας πούμε ε, προϊόντα. Εάν πρέπει ε, να ταξινομήσουμε το, το, το σύστημα αυτό ε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Εμείς βέβαια έχουμε ήδη προχωρήσει πάρα πολύ, γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε και σε ηγετική θέση και γι' αυτό θέλουμε να δίνουμε και τις δικές μας ιδέες όσον αφορά περαιτέρω ελέγχους, όσον αφορά ε, το ζήτημα της ε, οικονομίας και των ε, εταιριών. Όπως είπα και στην πρώτη μου παρουσίαση, ε, ξέρω ε, από την εμπειρία μου ότι οι εταιρείε έχουν ήδη εσωτερικές διαδικασίες οι οποίες ε, πάνε ακόμα παραπέρα και το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να το δούμε δε από πολλές πλευρές. Η μία από αυτές είναι ο έλεγχος των εξαγωγών, αλλά υπάρχουν και άλλα προγράμματα που μπορούν να οδηγήσουν σε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέλος, Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο σημαντικό να εστιάσουμε στα πιο ευαίσθητα θέματα όπως αυτά που ε, βλέπουμε σήμερα, αλλά θα πρέπει ε, να ε, δούμε και τα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από, ναι, από τις νέες βιομηχανίες και από τα εμπορεύματα τα οποία εξάγονται από άλλες χώρες πιο πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους εμπειρογνώμονες για αυτά που μας είπαν και είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι συνέχεια θα είναι πολύ καλή. Γιατί έτσι μπορούμε να συζητήσουμε για το μέλλον πώς θα χρησιμοποιήσουμε νομοθεσία. Νομοθεσία που περιμένουμε εδώ και πολύ καιρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω φέτος να την έχουμε και θα υπάρξει παρετέρω συνεργασία μεταξύ των δύο επιτροπών, δικαιωμάτων των ανθρώπων και ίντα δηλαδή, για το μέλλον του κανονισμού αυτού. Ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς πρέπει να φύγω γιατί αρχίζει η ίντα τώρα, οπότε σας εύχομαι καλή επιτυχία στο δεύτερο τμήμα. Thank you.

Vamos a tratar de empezar. Ας ε, αρχίσουμε με το δεύτερο τμήμα. Let's begin, please. Tenemos tenemos mucho de qué hablar en esta Σε αυτό το δεύτερο τμήμα έχουμε πολλά να πούμε και λίγο χρόνο. Γι' αυτό θα σας παρουσιάσω καταρχήν τους εμπειρογνώμονες που έχουμε μαζί μας εδώ σήμερα το πρωί για να συζητήσουμε τις επιπτώσεις επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ανάπτυξης όλων αυτών των ψηφιακών τεχνολογιών, των τεχνολογιών παρακολούθησης. Τι γίνεται με τη χρήση τους σε διάφορες χώρες του κόσμου και ποια είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να συζητήσουμε λοιπόν αυτό το θέμα έχουμε μαζί μας τον κύριο Φραν με εδώ αριστερά μου, ο οποίος ήταν ειδικό συζητητή των Ηνωμένων Εθνών για την πρόθεση και την προστασία του δικαιώματος ελευθερίας ε, γνώμης και έκφρασης. Είναι διευθυντής του κέντρου Ρόμπερτ Κέννεντι ε, στην Ευρώπη. Έχω επίση την κυρία Μαριάν Κνέρ, πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Επιστηλών στο Χίλτινσάιμ στην Γερμανία. Έχω τον κύριο Κένεθ Πέιτς που είναι υπεύθυνο ε, πολιτικών Privacy International είναι μια γνωστή οργάνωση και την κυρία Σαρά Μακίνα, η οποία είναι υπεύθυνη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο για το δίκαιο και την ψηφιακή ηθαγένεια κατά κάποιο τρόπο. Ο κύριος ε, Μίτσελσκι που είναι Διευθυντής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Γερμανία θα μας βοηθήσει στην συζήτηση αυτή. Έχετε 8 λεπτά μόνο για να μας μιλήσετε για τόσο περίπλοκα θέματα. Αλλά δυστυχώς βλέπετε σε αυτό το κοινοβούλιο πάντα έχουμε λίγο χρόνο. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Λαρή πρώτα απ' όλα και να ξέρετε ότι θα είμαι με το χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αυτή, κυρία Πρόεδρε, κυρία Συν Πρόεδρε Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να θέσουμε και πάλι ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για το παρόν και για το μέλλον. Θα είμαι σύντομος. Ο ιδιωτικό βίος και η ελευθερία έκφραση είναι δύο διαφορετικά δικαιώματα, αλλά πρέπει να τα κατανοήσουμε συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Και αυτό κάνω και εγώ με την έκθεσή μου. Δεν μπορεί κανείς να έχει ελευθερία εκφρασής πλήρω εάν συγχρόνως δεν έχει και την ε, εγγύηση για ιδιωτικό βίο. Αν δεν υπάρχει ιδιωτικός βίος, αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στο άτομο, είναι ένας εκφοβισμός, τον εμποδίζει να ασκήσει το δικαίωμά του ε, έκφραση ιδεών, ε, να τις γράψει, να τις σκεφτεί, να τις πει. Όλα αυτά επηρεάζουν τη δημοσιογραφία βέβαια. Υπάρχει η προστασία των πηγών και η προστασία του τύπου που είναι θεμελιώδη δικαιώματα αυτά για μια δημοκρατική ε, κοινωνία. Η ελευθερία έκφρασης διευκολύνει άλλα δικαιώματα, διευκολύνει την συμμετοχή των πολιτών, την άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών και αυτό γίνεται και μέσω του διαδικτύου. Τα ακούσαμε και πριν από λίγο όταν ο πληθυσμός της Τινησίας και της Αιγύπτου ύψωσαν τη φωνή τους. Ε, το μέλλον ήταν αβέβαιο αλλά οι φωνές τους ακούστηκαν και δικτατορίες 30 ε, ετής κατέρευσαν. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ότι αυτή η ελευθερία έκφραση είναι πολύ βασική. Τι γίνεται τώρα με την παρακολούθηση, ποια είναι τα προβλήματα. Η παρακολούθηση μπορεί να είναι νόμιμη όταν γίνεται στα πλαίσια του νόμου και της δημοκρατικής κοινωνίας. Ναι, το κράτος έχει την ευθύνη να προστατεύσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και την ασφάλεια των πολιτών. Και δεν συμφωνώ με τη συζήτηση εκείνη η οποία προσπαθεί να συνδέσει και να τα βάλει σε αντίφαση το ένα με το άλλο. Και τα δύο σε κάθε δημοκρατική δημοκρατία, σε κάθε δημοκρατική κοινωνία, συγγνώμη, πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ βασικό να ισχύσουμε την ασφάλεια, γιατί έτσι έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Αν λοιπόν η παρακολούθηση είναι απαραίτητη για να μπορεί κανείς να ερευνήσει εγκληματικέ δράσεις, τότε πρέπει να γίνεται. Φυσικά το σημερινό επιχείρημα είναι ότι με την ηλεκτρονική επικοινωνία, τα, την ψηφιακή τεχνολογία είναι πολύ δύσκολο να μπορεί κανείς να ελέγξει καλά τα πράγματα σε κάθε διαδικασία. Είναι διαδικαστικό το θέμα, αλλά τη διαδικασία πρέπει να την καθορίσουμε έτσι ώστε να υπάρχει ένα όργανο στο κράτος που να δίνει την εντολή, να μην είναι αυτό που κάνει την έρευνα να είναι χωριστά δηλαδή αυτός που δίνει την εντολή και αυτός που πραγματοποιεί την έρευνα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν χαθεί, είναι αλήθεια. Μερικά κοινοβούλια, οι κογκρέσα σε διάφορες ε, χώρες του κόσμου ελέγχουν τις δραστηριότητε αυτές, αλλά στην πραγματικότητα η διάσταση είναι τόσο τεράστια σήμερα που δεν έχουν την ικανότητα να το κάνουν. Έχουν δημιουργηθεί δικαστήρια για αυτό το σκοπό. Αλλά και πάλι είναι δικαστήρια τα οποία δίνουν ε, γενικές άδειες για παρακολούθηση, που σημαίνει ότι δεν εξυπηρετούν το στόχο προστασίας και ασφάλειας. Στη Γενέβη, κατά την εντολή μου, μπήκαμε σε μια συζήτηση ανάμεσα στην στοχευμένη παρακολούθηση και την γενική παρακολούθηση. Η γενική παρακολούθηση, εγώ είμαι πεπισμένος ότι όταν γίνεται σε μια άλλη χώρα είναι παραβίαση. Γιατί δεν υπάρχει περιορισμό στην άσκηση της εξουσίας αυτής. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εξισορρόπηση είναι πράγματα τέτοια που το κράτος ναι με τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά δεν πρέπει και να καταχράτε ποτέ της εξουσίας του στο όνομα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή της δημοκρατίας. Και επιμένω η ασφάλεια είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί αυτό σήμερα. Το Βέλγιο, για παράδειγμα, σήμερα περνάει από μια πολύ ειδική περίοδο και τα γεγονότα στο Σαρλί Εμπτό στο Παρίσι κατά πάσα πιθανότητα έχουν αλλάξει τη στάση της κοινή γνώμης ολόκληρη την Ευρώπη. Πιστεύω όμως η χρόνος ότι είναι σημαντικό να απαντάμε με συνέπεια, ενισχύοντας την δημοκρατία. Όταν είχαμε τα γεγονότα στο Όσλο, με τον κύριο Μπρέιβικ που σκότωσε νέα παιδιά, η απάντηση του Πρωθυπουργού της Νορβηγίας ήταν ότι πρέπει να φτιάξουμε μια μεγαλύτερη δημοκρατία, μια καλύτερη δημοκρατία, μια πιο ισχυρή δημοκρατία με συμμετοχή των πολιτών. Κατά κάποιο τρόπο αυτός είναι ο τρόπος για να ενισχύσουμε την ασφαλειά μας. Ποια είναι η βασική διάσταση Πρώτα απ' όλα, να αντιληφθούμε την ασφάλεια, τον ιδιωτικό βίο και την ελευθερία έκφραση ότι είναι τρία πράγματα που μπορούν να συνεπάρχουν. Δεύτερον, πρέπει να δούμε τις διαδικασίες να είναι δημοκρατικές, ανοιχτές, ώστε αν υπάρχει μηχανισμός παρακολούθησης να γίνεται μετά από άδεια και να ξέρουμε κατά πόσο είναι στοχευμένος ή γενικός. Γιατί πολλοί λένε εμείς σεβόμαστε τα δικαιώματα των ε, δικών μας ε, πολιτών, αλλά δεν το κάνουν όταν πρόκειται για χώρες αλλού. Αν όμως αρνηθούμε την οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αρνούμεθα και την οικονομικότητα, την οικουμενικότητα του διαδικτύου, η οποία πρέπει να παραμείνει. Είναι ζωτική σημασία. Πρέπει να προστατεύσουμε το διαδίκτυο. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό λοιπόν. Και τέλος, δεν μπορούμε να δεχτούμε την γενικευμένη παρακολούθηση σαν μια αναγκαιότητα πρέπει να είναι πάντα στοχευμένη με άδεια που έχει δοθεί δημοκρατικά και με έλεγχο των διαδικασιών από ένα άλλο κρατικό όργανο. Ιδεοδός θα πρέπει να συμμετέχουν και οργανώσεις ε, μη κυβερνητικές και σας συγχαίρω που τις καλέσατε σήμερα γιατί δεν μπορεί να γίνονται αντικείμενο εμπορίας ή εξαγωγών τα συστήματα αυτά παρακολούθησης. Πρέπει να τα δούμε πάντα χέρι-χέρι τα ανθρώπινα δικαιώματα με την ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που μας τα εξηγήσατε τόσο γρήγορα και τόσο ωραία. Θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς σε εσά. Τώρα η κυρία Μαριάν Κνόιερ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Συμπρόεδρε. Θα μιλήσω γερμανικά εάν είναι δυνατόν γιατί είναι η μητρική μου γλώσσα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να μιλήσω εδώ σήμερα. Στα επόμενα λεπτά θα ασχοληθώ με την ανάπτυξη και τα προβλήματα της ελευθερίας του διαδικτύου σε, σε ε, περιοριστικά καθεστώτα. σε καθεστώτα που, που περιορίζουν την χρήση του διαδικτύου. Και θα ήθελα να σας ε, καταδείξω πώς διαμορφώνεται η κατάσταση εμπειρικά. Και τέτοιες χώρες ε, τι μέτρα χρησιμοποιούν. Το διαδίκτυο είναι μια μεγάλη πρόκληση για αυτές τις ε, κυβερνήσεις. Αισθάνονται απλούμενες αυτές οι κυβερνήσεις από τέτοια καθεστώτα. Γιατί αυτό ε, επιτρέπει μια γρήγορη ε, επικοινωνία και αυτό αποτελεί εχθρό για τέτοια καθεστώτα. Äh, Regime auch das Internet, weil es natürlich auch ein... Τα πολιταρχικά λοιπόν καθεστώτα ε, βλέπουν ότι το διαδίκτυο ε, μπορεί να αποτελέσει και ένα εργαλείο για δικούς τους, την των δικών τους σκοπών. Άρα είναι λοιπόν ε, ε, διπλή η χρήση από πλευράς ε, των αυταρχικών καθεστώτων, των απολυταρχικών καθεστώτων. Έχουμε πολιταρχικά καθεστώτα που δεν επιτρέπουν ελευθερία του διαδικτύου και αυτό έχει ιδιαίτερα για την Ασία αλλά και στην Ευρασία και στην περιοχή της Κίνας, ναι, Βορειας Κορέας, Μιανμάρ, Σρια Λάνκα, Πακιστάν. Στην Ευρασία έχουμε τη Λευκορωσία, Τουρκμενιστάν, Ουσμπεκιστάν, αλλά και Ρωσία, Αζερβαϊτζάν, Καζακστάν. Και ύστερα έχουμε και την ε, Μπαχράιν, ε, Συρία, Αίγυπτο, ε, Τουρκία στη Μέση Ανατολή. Και η Τουρκία μας καταδεικνύει ότι όχι μόνο είναι πολυταρχικό καθεστώς, αλλά υπάρχουν και ευρεϊδικά καθεστώτα, τα οποία εμ, δρούν με τρόπο διτό. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι καταρχάς τα αυταρχικά καθεστώτα κατέχουν τεχνολογικά εξελιγμένες γνώσεις για να ελέγχουν το διαδίκτυο και για να ελέγχουν και την online επικοινωνία. Η τεχνολογική λοιπόν πρόοδος που επωφελεί τους χρήστες ε, έχει εφαρμογές και στις δυνατότητες παρακολούθησης. Αυτό το ακούσαμε και πριν από λίγο σε ό,τι αφορά τα τεχνολογικά στοιχεία. Αλλά διαπιστώνουμε άλλη μια εξέλιξη. Πέρα από την τεχνική αυτή μορφή της παρακολούθησης, τα τελευταία χρόνια έχει διαμορφωθεί μια τάση να επεκτείνονται νομικές ρυθμίσεις. Τι σημαίνει αυτό, ότι τα καθεστώτα πέρα από τον τεχνικό έλεγχο, ο οποίος ε, συνήθως εκφράζεται μέσω φίλτρων, μέσω ε, μπλοκαρίσματος ε, της μαζικής χρήσης, πλέον με νομικές ή με διοικητικές ρυθμίσεις προσπαθεί να εστιαστεί στο περιεχόμενο της επικοινωνίας online και αυτό επιτρέπει και τη δίωξη ατόμων κατά συνέπεια. Και γι' αυτό και αυξάνεται το ποσοστό δίωξη ατόμων σε τέτοια πολιταρχικά καθεστώτα. Έχουν αλλάξει λοιπόν τον τρόπο συμπεριφορά του ε, οι κυβερνήσει τέτοιου τύπου από μια αεραστεχνική, αν θέλετε, προσέγγιση που είχαν αρχικά και πλέον είναι αμυντική, εξελιγμένη η προσέγγιση τους και να αναφέρω κάποιες κατηγορίες τέτοιων μέτρων παρακολούθησης για να καταδείξω ποια είναι και η διάσταση, διάφορη διάφορε της παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Καταρχάς, έχουμε ε, θελούσια ε, κατασταλτικά μέτρα. Αυτό δεν είναι τίποτα καινούργιο στο διαδίκτυο, το ξέρουμε άλλωστε και από τα μέσα ενημέρωση, την ελευθεροτυπία, την ελευθερία έκφρασης γενικότερο. Ε, έχουμε σωματικές επιθέσεις, δολοφονίες, συλλήψεις δημοσιογράφων και έχουμε και την πρόσφατη ε, περίπτωση του Σαουδού σαν Σανταμπή. Αυτά συμβαίνουν ε, αλλά έχουμε κατά δεύτερον και σκληρούς ελέγχους και πάλι δεν θα κάνω διαχωρισμό μεταξύ τεχνικών μέσων και κατά δεύτερον ε, τεχνικών και διοικητικών ε, μέτρων. Τα τεχνικά μέτρα δεν θα επεκταθώ επ' αυτών γιατί ακούσατε ήδη τις πληροφορίες και φυσικά μπορούν να μπλοκαριστούν ολόκληρα δίκτυα, να γίνει λογοκρισία με φίλτρα, με, να μπλοκαριστούν διευθύνσεις IP ή για παράδειγμα λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναθετήσεις. Auf der Grundlage von schwarzen Listen gesucht werden. Diese τα νομικά τώρα μέτρα τα οποία μόλις ανέφερα αποσκοπούν στι δραστηριότητε ε, τις online και στα αντικείμενα επικοινωνίας. Όπως σας είπα, αυτές οι νομικές διατάξεις έχουν αυξηθεί, έχουν επεκταθεί τα τελευταία χρόνια. Ορίζονται αντικείμενα τα οποία θεωρούνται απαγορευμένα και απαγορεύονται. Όπως για παράδειγμα ο, χρησιμοποιούν την δικαιολογία της προστασίας της εθνικής ασφάλειας, της προστασίας της νεολαίας, των παιδιών, για τα κοινωνικά ήθη, για ε, την προστασία από πορνογραφικά υλικά, την προστασία από βλασφημία, την προσβολή θρησκευτικών συμβόλων, ε, προστασία από δηλώσεις κατά του κράτους και αυτό παλιά αγαπημένη δικαιολογία, ε, δυσφήμιση κτλ. Ο τομέας λοιπόν αυτός έχει πολύ επέκταση τα τελευταία χρόνια. Και τα διάφορα απαγορευμένα αντικείμενα έχουν μεγάλη ποικιλία. Με τέτοιε νομικέ λοιπόν διατάξει, αυτό που επιτυγχάνεται είναι το εξή. Στο εσωτερικό του εθνικού πλαισίου δημιουργείται μία νομική βάση για τέτοια καταστολή, για τέτοια δίωξη ατόμων, η οποία αποτελεί συνέπεια, και αυτό θεωρώ ότι είναι προβληματικό για μια ηθικά νομιμοποιημένη προάσπιση τέτοιων διατάξεων. Αυτό είναι προβληματικό πραγματικά. Η τρίτη δυνατότητα για τέτοια μέτρα αυστηρού ελέγχου βρίσκεται στον τομέα των ε, διοικητικών. Και εδώ τα τελευταία χρόνια λοιπόν είδαμε πως ε, έχει διαδοθεί αυτή η πρακτική και χρησιμοποιούνται κρατικές υπηρεσίες στον έλεγχο του διαδικτύου. Δίνεται λοιπόν και εδώ μια νόμιμη δικαιολογία για τον έλεγχο, για παράδειγμα, δηλώσεων που στρέφονται κατά του κράτους, επιθεωρητές, πολι... Ε, αστυνομία στο διαδίκτυο ή σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, την ενδεχόμενη καταχώρηση, η σε οτι αφορα για παραδειγμα την ενεχομενη καταχωρηση η οποια και αυτή επιτρέπει με τη σειρά της ως διοικητικό μέτρο τον έλεγχο. Κατά τρίτον, βλέπω ότι υπάρχει και παρατηρεί κανεί τη δυνατότητα ήπιων μέτρων. Πέρα από τα σκληρά μέτρα υπάρχουν και τα ήπια μέτρα παρακολούθησης. Τα απολυταρχικά καθεστώτα όλο και πιο πολύ χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για τον σκοπό της νομιμοποίησης του καθεστώτος τους. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις ή απολυταρχικές το χρησιμοποιούν, αξιοποιούν το ίντερνετ σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, το e-government, την ηλεκτρονική κυβέρνηση ή participation, ηλεκτρονική συμμετοχή. Τα χρησιμοποιούν λοιπόν αυτά για να νομιμοποιηθούν έναντι των λαών τους, για να ζητήσουν υποστήριξη. Προγράμματα, τα προγράμματα e-government, αυτό το βλέπουμε και στα προγράμματα τα σχετικά του ΟΗΕ, υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα τα οποία προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες στους πολίτες τους προκειμένου να προσποιηθούν ότι υπάρχει διαφάνεια και ισότητα δικαιοσύνη. Και το ίδιο συμβαίνει και με προγράμματα e-participation. Για παράδειγμα, τα blog, σελίδες στο διαδίκτυο οι οποίες υποτίθεται ότι προσφέρουν ε, τη δυνατότητα στους πολίτες να μιλούν, να συνομιλούν με τα μέλη της τοπικής τους κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και αυτό πάλι δίνει μια εντύπωση α, ε, συμμετοχής. Τέτοιες λοιπόν χώρες που κάνουν τέτοιες ε, προσωμιώσεις είναι το Μπαχρέν, Σιγκαπούρη, Καζακστάν, Εκεί λοιπόν υπάρχει ήδη μεγάλη παράδοση και εμπειρία. Τέλος, τέτοιες, ε, τέτοια πολιταρχικά καθεστώτα μπορούν να κάνουν και προπαγάνδα μέσω του διαδικτύου. Αυτό γίνεται όλο και πιο συχνά. Αυτές είναι οι μέθοδοι, οι νέες μέθοδοι που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια για την ε, Ενεργεί τέτοια στάση των απολυταρχικών καθεστώτων με... είναι ένας τρόπος με τον οποίο να ε, εκμεταλλεύονται το διαδικτύο για να ενισχύσουν την νομιμότητά τους. Αυτό έχει με τη σειρά του επιρροή στην επίθεση στο μεμονωμένο άτομα αλλά έχει και συνέπειες ε, για τον κοινωνικό έλεγχο σε ό,τι αφορά τα πολυταρχικά αυτά καθεστώτα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος και τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος Kenneth Page από την Privacy International. Σας ευχαριστώ. Υπεύθυνος πολιτικών. Κύριοι Πρόεδροι, αξιότιμα μέλη, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό να βλέπουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα σε σχέση με τις ε, σύγχρονες ε, τεχνολογίες να βρίσκονται τόσο ψηλά ε, στο θεματολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάρα πολλές οι χώρες οι οποίες δίνουν τέτοιου είδους εξοπλισμό σε πάρα πολλές χώρες του είναι θέμα το οποίο εμείς έχουμε ήδη ε, σημειώσει και ε, ε, στη συνεργασία και με άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Εμείς καλούμε τις κυβερνήσεις να επικαιροποιήσουν, να εξυγχρονίζουν την πολιτική εξαγωγών ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να δούμε ότι αυτού του είδους ε, το εμπόριο δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα φτάνοντας μέχρι βασανισμό, εκτοπισμό ε, εξορία, ε, φυλακισμό ανθρώπων ε, και αναφερόμαστε σε ακτιβιστές, σε αντιφρονούντες, σε δημοσιογράφους κτλ. Υπάρχει μάλιστα και ένα anti-intrusion software το οποίο συχνά χρησιμοποιείται έτσι ώστε να, έτσι ώστε να σπάσει τα antivirus συστήματα τα οποία μπορεί να έχουν εγκατασταθεί στους υπολογιστές. Ε, εμείς ε, ξέρουμε ότι, ε, σε κάθε, ότι μετά από κάθε μεταβίβαση εμπορική μπορεί να δημιουργηθούν νέες σειρές προβλημάτων τα οποία δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Τα τελευταία χρόνια έχει, είναι πολλές χώρες αυτές οι οποίες έχουν δημιουργήσει μεγαλύτερες ε, ε, μεγαλύτερα ακόμα προβλήματα, έχουν προκαλέσει προβλήματα μεγαλύτερα ακόμα ε, σε αντιφρονούντες σε χώρες όπως το Μπαχρέιν ή όπως το Βιετνάμ. Και ξέρουμε ότι οι γαλλικές εταιρείες έχουν επανειλημμένα πουλήσει υλικό στην Σύρια. Επίσης στην Κεντρική Ασία σε πάρα πολλές χώρες έχει πολιθεί υλικό το οποίο έχει δημιουργήσει προβλήματα σε αντιφρονούντες, στο Μπαχρέιν και αλλού αλλού. Ε, επίσης γνωρίζουμε ότι στο Μπαγκλαντές ε, οι αστυνομικές δυνάμεις ε, έχουν παρακολουθήσει παράνομα πολλές φορές αντιφρονούντες ή αντιτιθέμενους στην κυβέρνηση μέσω παρακολούθησης ή αμπλοκαρίσματος των κινητών τους τηλεφώνων. Ε, επίσης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένα έχουν ε, καταγραφεί και καταγγελθεί τέτοιου είδους παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Βλέπουμε ότι είναι ανησυχητική όμως η αύξηση τέτοιων κρουσμάτων παντού. Έχουμε πλέον συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι το Υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου προσπαθεί να αγοράσει υλικό καταστολής ε, έτσι ώστε να παρακολουθεί όλα τα ε, κοινωνικά δίκτυα. Ε, η Αραβική Άνοιξη επίσης έδειξε ότι αυτές οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν οποιοδήποτε μέσο έτσι ώστε να μπορέσουν να καταστήλουν την συνεννόηση και την επικοινωνία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει εμπάργο ε, για τεχνολογίες οι οποίες ε, χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των πολιτών. Το 2014 έχουμε αποδείξεις ότι η Ιταλική εταιρεία Hacking Team χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να στοχοποιηθούν δημοσιογράφοι με έδρα της Ηνωμένε Πολιτείες που εργάζονταν για ανεξάρτητα αιθιοπικά μέσα ενημέρωση. Το 2012 είδε τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε έτσι ώστε να στοχοποιηθούν ε, μαροκινοί πολίτες ε, του Media Group Mam Fakins και επίσης αυτού του είδους ε, ε, πανευατικό λογισμικό μπορεί να αντιγράψει files ε, από οποιαδήποτε, από μηχάνημα το οποίο έχει προσβληθεί. Μπορεί επίσης να καταγράψει τις κλήσεις μέσω Skype, τα email, τα, τα μηνύματα καθώς επίσης και να σπάσει κωδικούς. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει και να ανοίξει μόνο του μικρόφωνα και κάμερες. Ε, τα ε, hacking, η hacking team, η εταιρεία hacking team διαφημίζει το προϊόν της ε, ως δυνάμενο να στοχοποιήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων. Αυτή η εταιρεία όπως και πάρα πολλές άλλες λέει βεβαίως ότι πουλάει σε τελικό χρήστη το, σε, σε χρήστες που είναι οι τελικοί χρήστες και είναι κυβερνήσεις. Ε, αυτό θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά ε, υπόψη μας. Βεβαίω ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και να ακούσουμε τις μη κυβερνητικέ ε, οργανώσεις και αυτά που έχουν να μας πούν ε, για τα θέματα αυτά. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφέρθηκε σε τέτοια προβλήματα τα οποία σχετίζονται με την πολιτική εξαγωγών. Τον προηγούμενο Νοέμβριο αναφέρθηκε συγκεκριμένα μέσω εκθέσεως ότι τέτοιου είδους υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να εντοπιστεί για τον εντοπισμό, την υποκλοπή ε, και την παρακολούθηση τηλεφωνικών ε, επικοινωνιών. Ε, εμείς ε, πιστεύουμε ότι η ίδια η πολιτική εμπορίου ε, θα πρέπει να συμμορφώνεται προς κάποιες αρχές όπως είναι η ασφάλεια, όπως είναι η διαφάνεια, όπως είναι η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ο έλεγχος των εξαγωγών δεν είναι ένα εργαλείο έτσι ώστε να δημιουργηθούν προβλήματα στις εξαγωγικές εταιρείε, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν με, να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο σωστό έτσι ώστε ε, να ε, ε, προστατευτεί ε, ο πολίτης. Ε, η κύρια πρόκληση είναι να βρούμε τον σωστό ε, μέσο όρο, να βρούμε τον σωστό τρόπο έτσι ώστε να μην απαγορευτούν οι εξαγωγές από τη μία αλλά και να μην δημιουργηθούν τα εργαλεία τα οποία θα αποτελέσουν επιπλέον εργαλείο στην καταστολή και στην παρακολούθηση. Ο στόχος ε, είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα ε, τα οποία θα έχουν δημιουργηθεί με συγκεκριμένο και στοχευμένο τρόπο έτσι ώστε ε, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καλή λεγόμενη παρακολούθηση και σίγουρα όχι την μαζική παρακολούθηση. Η κοινωνία των πολιτών μπορεί σημαντικά να συμβάλλει στον τομέα αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση οπωσδήποτε θα πρέπει να λάβει υπόψη της την διαμόρφωση νέων μηχανισμών όσον αφορά τον έλεγχο ε, των εξαγωγών και την γενικότερη πολιτική εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κυρίως το θέμα του τελικού χρήστη και του πώς καθορίζεται ο τελικός αυτός ε, χρήστης η Αραβική Άνοιξη μας έχει δείξει ότι είναι πολλές οι κυβερνήσεις οι οποίες χρησιμοποιούν την ε, τεχνολογία η οποία πωλείται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του δυτικού κόσμου έτσι ώστε ε, να παρακολουθήσουν, να υποκλέψουν ε, και να καταστήλουν. Ε, ε, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να ξαναβρούμε, να ξαναδούμε και τις 21, τα 21 στοιχεία όσον αφορά τις εξαγωγικές άδειες για υλικό παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων κυρίως όσον αφορά χώρες όπως την Αιθιοπία, το Τσάτ, το Τουρκμενιστάν και η Εμένη. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Πέιτζ. Και κυρία Σάρα Κίνε, ερευνήτρια. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να συμμετάσχω σήμερα στην ακρόαση αυτή. Είμαι ανώτατη νομική σύμβουλος της Citizen Lab. Η οργάνωσή μας έχει ετοιμάσει τεκμηρίωση το τελευταίο καιρό σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε χρησιμοποιήσει πραγματογνωμοσύνη, νομική και τεχνολογική. Έχουμε δει ότι κίνδυνο ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις ψηφιακές τεχνολογίες υπερβάλλονται μερικές φορές στις κοινωνίες στις οποίες βρισκόμαστε. Όλοι μας είμαστε δικτυωμένοι, αλλά λίγοι έχουν ασφάλεια στη δικτύωση αυτή και λίγοι από τους προνομιούχους χρησιμοποιούν και την κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει περισσότερος έλεγχος για όλον τον πληθυσμό ε, στις χώρες μας και εκτός. Οι απειλές δεν έχουν σύνδεση μόνο με την κυβέρνηση. Υπάρχουν ε, έρευνες που έχει κάνει το Citizen Lab που δείχνουν τις ψηφιακές απειλές. Έχουμε τέσσερα χρόνια τώρα κάνει μελέτες και έχουμε ετοιμάσει έκθεση όπου θα βρείτε πολλές λεπτομέρειες. Πρόκειται για την έκθεσή μας που ονομάζεται Communities at Risk. Το κακόβουλο λογισμικό όταν χρησιμοποιείται, ε, χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν γνωρίζουμε πάντα. Θα έπρεπε να είναι προτερότητά μας να έχουμε απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα και να έχουμε περισσότερη διαφάνεια. Έρχομαι στις συστάσεις. Τι ξέρουμε. Πρώτον, στον ψηφιακό κόσμο οι κοινωνίες των πολιτών και οργανώσεις τους έχουν τις, αντιμετωπίσει τις ίδιες απειλές όπως και ιδιωτικό τομέα και κυβέρνηση, αλλά είναι λιγότερο εξοπλισμένοι. Βλέπουμε ότι πολλοί ε, πλήττουν την κοινωνία των πολιτών, το κάνουν και με επιχειρήσεις και με κυβερνήσεις και στη μελέτη μας είδαμε ότι πολλοί από αυτούς είχαν ε, συνδέσεις με αυτούς που προχωρούν στις απειλές. Έπειτα, η τεχνολογική διάσταση δεν είναι τόσο σημαντική στα κακόβουλα λογισμικά. Το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζουν το στόχο τους καλά. Οι, τα περισσότερα κομπιούτερ που εξετάσαμε δεν είχαν προβλήματα. Αυτό που διαπιστώσαμε ήταν ε, ότι σε πολύ λίγο, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μπορούσαν να προχωρήσουν οι απειλές αυτές. Τι επιπτώσεις έχουν ε, αυτά, η χρησιμοποίηση δηλαδή κακόβουλων λογιστικών. Είτε πρόκειται για περίπλοκη τεχνολογία, είτε πρόκειται για απλή, η ζημιά που γίνεται είναι ίδια, γιατί μπορούν να μπουν μέσα σε φακέλους, όταν ε, έχουμε να κάνουμε με πιο περίπλοκα λογισμικά παρίσδησης, βλέπουμε ότι ο τρόπος να τα αντιμετωπίσουμε είναι ο έλεγχος των εξαγωγών. Οι ψηφιακές επιθέσεις στην κοινωνία των πολιτών, στις κυβερνήσεις και άλλες οργανώσεις είναι κάτι συνεχιζόμενο. Γίνεται παντού και πάντα. Η επιμονή αυτή δείχνει ότι είναι ε, πολύ αποφασισμένος αυτός που επιτίθεται να πετύχει το στόχο του. Οι ψηφιακές απειλές υπονομεύουν τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην επικοινωνία τους πάρα πολύ σημαντικά και φτάνει μερικές φορές στη ζημιά και στην ατομική ασφάλεια. Οι απειλές αυτές υπονομεύουν λοιπόν και την αποτελεσματικότητα των οργανώσεων γιατί δεν μπορούν να πετύχουν το στόχο τους. Υπάρχουν βέβαια και οικονομικά προβλήματα. Οι υποδομές και επαγγελματίες είναι αυτό που χρειάζεται για να αντιμετωπιστούν οι απειλές αυτές. Και οι ψυχολογικές είναι οι συνέπειες. Τα ψηφιακά μέσα, το Skype ή άλλα, around the world, but are known to have been targeted for government compromise in the past.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 περιέγραψε τι συνέβη με το λογαριασμό του Skype. Υπήρχε παρεμβολή σε αυτόν και ήταν πολύ ταραγμένη για μέρες. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις οι ψηφιακές ε, τέτοιες παρεμβολές επηρεάζουν γιατί την αποστολή των ε, κοινωνικών οργανώσεων αλλά και τα άτομα ατομικά.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 ε, περιορίζουν τα δικαιώματα και τον τρόπο λειτουργίας των θυμάτων. Είναι πράγματα τα οποία συζητιούνται πολλές φορές στις χώρες που υποφέρουν από αυτά. Θα πρέπει να υπάρχει ένας ε, συμβασμός η μελέτες που έχουν γίνει έχουν δείξει ότι είναι στο Ταραλσαλάμα και αλλού τέτοιες οργανώσεις που επιτίθενται Κάποια άλλα, κάποια λόγια για τις προσπάθειες για διαφάνεια. Τα σχετικά προϊόντα. Στην παρούσα φάση δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε την ε, ορατότητά τους από τη βάση αυτή. Ποιοι μηχανισμοί λοιπόν μας θα επιτρέψουν να υπάρχει αυτή η διαφάνεια, αυτή η ορατότητα. Οι εσωτερικοί ε, κανονισμοί των εταιριών είναι ένα ε, θέμα για το οποίο επίσης δεν γνωρίζουμε πολλά. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε μέτρα κοινωνικής ευθύνης και ότι τα, οι σχετικέ ε, ρυθμίσει θα είναι ανοιχτέ στον ε, δημόσιο διάλογο. Χρειάζεται πιο πολλέ πληροφορίε για τι ε, αλυσίδε διανομή, για την μεταφορά τεχνολογία. Και πολλέ εταιρείε διπλή τεχνολογία ε, υπολογίζουν ότι υπάρχει απόσταση από το προϊόν όλο και πιο μεγάλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο πολλέ πληροφορίες για τις αλυσίδες αυτές διανομής και να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή για να υπάρχει και καλύτερη λογοδοσία. Τέλος, ποιοι πριάζονται. Ξέρουμε ότι η κοινωνία των πολιτών αποτελεί το στόχαστρο και πολλά ακόμα θα πρέπει να μάθουμε και πολλά θα πρέπει να κάνουμε για να αποκαλύψουμε τέτοιες ε, ε, παρισδήσεις. Σε ό,τι αφορά τις συστάσεις, από ό,τι φαίνεται στον κυβερνό χώρο, έχουν ε, αυξηθεί οι γνώσεις μας, αλλά βρισκόμαστε σε μια φάση που μπορούμε να αποτρέψουμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Χρειαζόμαστε πιο καλή τεκμηρίωση των περιστατικών αυτών. Να συλλέξουμε δεδομένα για ανησυχίες, για σεβασμό της, του απορρίτου. Τα εμπορικά μέτρα, όπως η έλεγχη για παράδειγμα εξαγωγών, αποτελούν έναν τρόπο να ελέγξουμε τις ψηφιακές απειλές, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται και από πολιτική υποστήριξη, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε σωστά τις ε, σχετικέ απειλές. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε στο ότι κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να είναι εκτός των ορίων της κατασκοπίας και της ψηφιακής στοχοθεσίας. Θα πρέπει να βρούμε μια εντολή στα πλαίσια του ΟΗΕ για να χρησιμοποιήσουμε ε, το... ό,τι δυνατότητα έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την ψηφιακή απειλή. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο πολλές δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τις αστάθειες για την ψηφιακή ασφάλεια. Θα πρέπει να σκεφτούμε τα σχετικά πρότυπα που ισχύουν για το hardware και το software από τον μέσο άνθρωπο για να υπάρχει λύση εξ αρχής. Θα πρέπει να κοιτάξουμε λύσεις ε, για την ιδιωτική σφαίρα, για την κρυπτογράφηση, επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία δεν θα υπονομεύουν ε, την ασφάλεια και την ιδιωτική σφαίρα. Σε ό,τι αφορά την κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συνεχίζουμε να δίνουμε απαντήσεις στα ερωτήματα και τις ανησυχίες. Στο ιδιωτικό τομέα θα πρέπει να υπάρχει ε, μια κανονική ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σαν κάτι το οποίο ε, υπάγεται στις ε, όρους της αγοράς. Είναι λοιπόν ένα σημαντικό τμήμα αυτό και τέλος η έρευνα και τα εργαλεία για την ασφάλεια θα πρέπει να λαμβάνουν κίνητρα για να υπάρχουν επενδύσεις σε λύσεις που θα προστατεύουν την κοινωνία από τέτοιες Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν ποια νομοθεσία χρειάζεται για να προστατεύει το κοινό και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρακολουθούν την ανάπτυξη της αγοράς για εργαλεία τα οποία θα υπονομεύουν την ασφάλεια σε τέτοιο επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μακίνε. Συγγνώμη για την διακοπή. Συγγνώμη και από τους διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος, αν δυσκολεύτηκαν. Ίσως να φταίω εγώ. Γιατί εγώ ζήτησα από τους προσκεκλημένους να μιλήσουν σε 8 λεπτά και βέβαια είχαν τόσα πολλά να μας πούν. Είναι άνθρωποι που έχουν εμπειρία και ξέρουν ότι πρέπει να μιλάνε πιο αργά για να μπορεί κάποιος να τους μεταφράσει. Ευχαριστώ πάντως τους διερμηνείς που έτσι αλλιώς είναι εξαίρετοι επαγγελματίες. Ευχαριστώ και την κυρία Μακιούν για την εξαίρετη παρουσίασή της. Και τώρα, τελευταία σχόλια. Θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Human Rights Watch, τον κύριο, στη Γερμανία τον κύριο Μισάλσκι. Σας ευχαριστώ. Θα χρησιμοποιήσω τη μητρική μου γλώσσα αν ε, ε συμφωνείτε. Ίσως κάποια στιγμή αναφέρω και κάτι στα αγγλικά, μια σκηνική λίγου αφράγκα. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να εκφράσω καλύτερα στα γερμανικά. Καταρχάς να πω ότι με εντυπωσίασε ιδιαίτερα το πρώτο πάνελ σε ό,τι αφορά τον έλεγχο εξαγωγών. Το ότι υπήρχαν τόσο πολλά άτομα εδώ που δεν έφταναν καν οι θέσεις. Τώρα λοιπόν που μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχει μειωθεί η προσέλευση. Ελπίζω αυτό να σχετίζεται πιο πολύ με κάποια άλλη πιο σημαντική εκδήλωση και να μην είναι ένα σύμπτωμα, ένας κακός ιονός αυτά που, για αυτά που συζητάμε εδώ σήμερα. Στο πάνω λοιπόν αυτό επικρατεί μεγάλη συμφωνία γενικότερα για το πόσο σημαντικά είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές ε, τεχνολογίας ε, παρακολούθησης. Αυτό δεν ήταν ε, το ίδιο στο πρώτο πάνελ. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να εστιάσω κυρίως στα σχόλια που έχω να κάνω για το πρώτο πάνελ. Όχι μόνο σε αυτό βέβαια. Ήταν το ασφαλώς αυτό που είπε ο κύριος Κρίστιαν Χόιχερτ και η ερμηνεία που δίνει στην κερατομία και στις τεχνολογίες. Αυτή η ερμηνεία πραγματικά μου υπενθύμησε σκοτεινές στιγμές του 20ου αιώνα. Όταν η κοινοτομία της τεχνολογίας ήταν πάνω από όλα και ο αντίκτυπος του ανθρώπινου δικαιώματο δεν έπαιζε κανένα απολύτως ρόλο. Και καταλαβαίνω εν μέρει αυτά που είπε και ο κύριος Ντέους, αλλά ίσως θα ήθελα να το θέσω υπό, υπό διαφορετικό πρίσμα. Να δώσω κάποια παραδείγματα για αυτά που έκανε το Human Rights Watch τα τελευταία χρόνια στην Αίγυπτο. Όταν ε, η Αραβική Άνοιξη πρώτο ξεκίνησε και έπεσε το καθεστώς του Μουμπάρακ, ε, μια γερμανική ομάδα της τηλεόρασης βρέθηκε στο Κάιρο και βρήκε μια επιστολή μιας γερμανικής ε, εταιρείας παρακολούθησης όπου η εταιρεία αυτή πρόσφερε να αναλάβει την παρακολούθηση των αντιφρονούντων για το Μουμπάρακ. Λίγο πολύ η επιστολή έλεγε ότι «Α, έχετε ένα πρόβλημα με την επαναστασή σας, εμείς θα φροντίσουμε το πρόβλημα αυτό να επιληθεί». Τώρα, ο, το καθεστώς Σίση έκανε μία δημόσια διαγωνισμό με σκοπό να βρει να αγοράσει ευρωπαϊκή ευρωπαϊκό, ε, ευρωπαϊκή τεχνολογία παρακολούθησης. Γιατί είναι πιο αποτελεσματική η ευρωπαϊκή τεχνολογία μετά την ε, σφαγή Tianmen, ε, το καθεστώς της ΣΥΣΥ έκανε την πιο αποτελεσματική μαζική, μαζικές εκτελέσεις. στρατιωτική, αστυνομική παρακολούθηση φροντίζουν προκειμένου να φυλακίζονται, να δολοφονείται οποιαδήποτε αντιπαράθεση και αντιπολίτευση. Παρ' όλα αυτά, χωρίς ε, να ντρέπεται ξεδιάντροπα να ζητά ευρωπαϊκή τεχνολογία. Ένα άλλο παράδειγμα, η Συρία. Το 2011 για πρώτη φορά τα κράτη-μέλη φρόντισαν οι εξαγωγές ε, παρακολούθησης, τεχνολογίες παρακολούθησης προς το καθεστώς Αστάτ να ε, ελέγχονται και να σταματήσουν. Το 2011 στο Μπαχρέιν συνεχίζονται οι εξαγωγές κατά πάσα πιθανότητα ακόμα σήμερα. Γιατί ε, φυλακίζονται οι προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι τελικά έχουν συλληφθεί βάσει τεχνολογιών παρακολούθησης. Ε, περνάνε από, βασανιστήρια, συλλαμβάνονται οι οικογένειές τους και δεν μπορούν να... Ε, άλλοι εξορίζονται, άλλοι δεν μπορούν να βγουν από τη χώρα. Η Αιθιοπία. Η Αιθιοπία είναι μια χώρα που αξιοποιεί ε, πολύ εκτεταμένα και με πολύ ευθύ τρόπο την Ευρωπαϊκή Τεχνολογία Παρακολούθησης. Η Human Rights Watch ε, δημοσίευσε το 2011 μια εκτενέστατη έκθεση όπου διαπιστώνεται πως οι αντιφρονούντες, ε, οι δημοσιογράφοι ε, διώκονται με την χρήση ευρωπαϊκής τεχνολογίας, πώς φυλακίζονται, βασανίζονται, εξαφανίζονται, εκτελούνται. Και ακόμα και στην εξορία, με τη βοήθεια του λογισμικού τη τεχνολογία αυτή, παρακολουθούνται ακόμα και στην εξορία. Στην Νορβηγία, για παράδειγμα, υπάρχει μια ομάδα η οποία παρακολουθεί άτομα τα οποία έχουν διωχθεί από την Αίγυπτο. Και ασκείται πίεση στην οικογένεια, για παράδειγμα, του αντιφρονούντος στην Νορβηγία, στην οικογένειά του στην Αιγυπτό, προκειμένου να μην εκφράζει ελεύθερα την ε, γνώμη του, την απόψή του, γιατί αλλιώς θα απειληθεί η οικογένειά του. Δυσίωνο και σκοτεινό. Και αυτή η τεχνολογία είναι μη αντιληπτή. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε ότι για παράδειγμα είναι πάρα πολύ ευφύης τεχνολογία. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χρησιμοποιείτε τη τηλέφωνό σας, τον υπολογιστή σας. Και Γι' αυτό είναι τόσο επικίνδυνη στα χέρια των λάθο ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω την επιχειρηματολογία των προηγούμενων ομιλητών. Προφανώ ε, πρέπει να υπάρχει καινοτομία, να υπάρχει επιστημονική πρόοδο. Θα είναι αστείο και ανόητο να υποστηρίξουμε το αντίθετο. Όχι ει βάρο ανθρώπινων ζώων όμω, ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όπου σε τέτοιε ακραίε περιπτώσει τι οποίε μόλι ανέφερα. Και γι' αυτό λοιπόν είναι τελείως παρανοϊκό το, οποίο, το ότι ο κύριος Χόχε πρότεινε ως εκπρόσωπος μιας ομάδας η οποία ε, δραστηριοποιείται από τη δεκαετία του 80 για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτά. Χρειάζεται κάποια απόσταση διαφορετικά. Ήταν αυτά που μας είπε ο κύριος Νορτέους. Είναι φυσικά κατανοητό ότι όλοι έχουμε συμφέροντα, πόσο μάλλον και η βιομηχανία. Όλοι θέλουμε να προωθηθούμε, να υπάρξει πρόοδο, να υπάρχουν θέσει απασχόληση, ανταγωνισμό. Αλλά και εδώ υπάρχουν όρια. Και αν ε, τα πάρετε στα σοβαρά αυτά που μόλι σα περιέγραψα και υποθέτω θα τα πάρετε στα σοβαρά. Θα ζητήσετε αυθορύθμιση αλλά δεν θα έχετε και αντίρρηση να ελεγχθούν οι εξαγωγές. Αν υπάρχουν οποιαδήποτε ε, ερωτήματα, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο σε κάθε ε, Υπουργείο Εξωτερικών και να ρωτήσετε κατά πόσον ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την ανεμοθεσία για τον έλεγχο των εξαγωγών ή μήπως υπάρχουν κάποια προβλήματα για τα οποία θα πρέπει να μεριμνήσουμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι πέρα από την ανταγωνιστικότητα, η οποία σύμφωνη χρειάζεται προκειμένου η τεχνολογία αυτή να μην παράγεται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν άλλο, άλλα πρότυπα και να μην έχουν προτέρημα αυτές οι χώρες. Θεωρώ όμως ότι το επόμενο βήμα το οποίο θα πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει μια παγκόσμια ρύθμιση σε επίπεδο ΟΗΕ. Και εκεί νομίζω θα λυθεί και το θέμα τη ανταγωνιστικότητα το οποίο τίθεται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μιτσάλσκι. Θα δώσω τώρα το λόγο στου ευρωβουλευτέ. Και μετά στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση. Είναι εδώ η κυρία Νιέβες Φερνάντε, σωστά. Δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε για διάφορους λόγους να μην πάρει το λόγο. Έχουμε όμως την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Συνεπώς, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βάιντεν Χόλσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος ε, Μιχάλσκι, πολύ φοβάμαι ότι έχετε απόλυτα δίκιο με την παρατήρηση που κάνατε ότι κατά τη δεύτερο ήμιση του πάνελ είναι πολύ πιο μειωμένη η προσέλευση του κόσμου, γιατί αυτό είναι ένα γενικό φαινόμενο. Μειώνεται η προσέλευση όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι τα δύο αυτά θέματα, οι δύο αυτές πτυχές εξετάζονται από κοινού. Και εντάξει, ίσως το πρώτο τμήμα ήταν πιο πολύ παριστάμενοι. ακούγοντας τους διάφορους συναδέλφους, ε, ε, ε, δημιουργείται μια αίσθηση αδυναμίας, πλήρους αδυναμίας. Αν σκεφτούμε όλα αυτά που μας είπατε για τις τεχνικές δυνατότητες που υπάρχουν, πριν από δύο-τρία χρόνια νομίζω ότι συζητούσαμε και θα είχαμε συζητήσει πολύ πιο αισιόδοξα όλα αυτές τις τεχνικές δυνατότητες, αλλά και την αμιμότητα Θυμάμαι μια συζήτηση που είχαμε την τελευταία, στην τελευταία αλλαμέλεια στο Στρασβούργο όπου μιλήσαμε για την κατάσταση στην Αίγυπτο και όπου ακούσαμε από διάφορους συναδέλφους ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη σταθερότητα και για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτή τη σταθερότητα θα πρέπει προσωρινά ίσως να κάνουμε και τα μάτια για τέτοια ζητήματα. Θα ήθελα να θέσω τη διάσταση του διεθνούς εμπορίου, γιατί μόνο μέσω του έλεγχου των εξαγωγών μπορούμε να έχουμε οποιοδήποτε έλεγχο και να μην είμαστε εντελώ αδύναμοι. Είναι λοιπόν θετικό και εντραντικό το γεγονός ότι ήταν πολλοί συναδελφοί που ήλθαν στο πρώτο πάνελ και ε, εκφράστηκαν. Νομίζω ότι ένα από τα σημαντικά σημεία τα οποία θα πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε είναι το τι κάνουμε εδώ στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να κάνουμε ελέγχου εξαγωγών και εμεί να υποκρινόμαστε ότι στο εσωτερικό όλα πάνε καλά. Ο κύριο Λαρούι μίλησε για βασικές αρχές ε, σκεφτόμενος ε, διάφορες, ε, διάφορα περιστατικά για την, ε, τα προσωπικά δεδομένα, για τη χρήση βίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε και ενδεχομένως μήπως κάποια πράγματα υπερβαίνουν αυτά που έχουμε πετύχει στην ε, δυτική κοινωνία. Ε, Ευχαριστούμε. Η κυρία Λόκμπιλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ όλους σας για τις πολύ καλές παρεμβάσεις. Μία ερώτηση θα ήθελα να απευθύνω προς την κυρία καθηγητρία Κνόερ. Με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια παρουσιάσατε πώς τα πολυταρχικά καθεστώτα χρησιμοποιούν αυτές τις ψηφιακές τεχνολογίες. Και εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα λοιπόν ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρειαζόμαστε μια λεπτομερή λίστα, ένα λεπτομερή κατάλογο που θα περιγράφει πώς έχει η κατάσταση στις χώρες αυτές προκειμένου ενδεχομένω να αποκλειστεί τέτοια τεχνολογία λογοκρισίας, τεχνολογία που επιτρέπει δίωξη ατόμων από ενδεχόμενες εξαγωγές. Να απαγορευτούν οι εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, μέσω τέτοιων εταιριών που έχουν έντρα σε χώρες αυτές. Έχετε λοιπόν κάποια πρόταση και είναι Κρίμα που δεν είναι εδώ μαζί μας πλέον η Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω και σας κάτι, γιατί ο πρόσωπος του πρώτου πανέλ είπε ότι είναι δύσκολο να αποφασίσουμε τι είδους τεχνολογία θα πρέπει να απαγορεύεται όταν μιλάμε για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν όμως κοιτάξουμε τους προορισμούς της χώρας στις οποίες δεν θα πρέπει να εξαγάγεται τεχνολογία, ίσως τα πράγματα να είναι πιο απλά. Αν, για παράδειγμα, λέγαμε ότι υπάρχουν απολυταρχικά καθεστώτα, θα μπορούσαμε να αποφασίσουμε ότι δεν εξαγάγουμε σε αυτές τις χώρες. Μία ερώτηση για το Human Rights Watch. Μία ερώτηση. Μας είπατε ότι θα πρέπει οι οργανώσεις να προστατευτούν μέσω συνεχιζόμενη εκπαίδευση στι αναπτυσσόμενε τεχνολογίε. Γιατί ε, εξειδικεύονται και οι απολυτρικές κυβερνήσει. Υπάρχουν λοιπόν κάποιε προσφορέ ε, διοργάνωση τέτοιων εκπαιδεύσεων, τέτοιων προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω αν υπάρχει ζήτηση, μεγαλύτερη ζήτηση για τέτοια προγράμματα ή μήπως πρέπει για προγράμματα που δεν αξιοποιούνται. Και προς την κύριο Page θα ήθελα να σας κάνω κάποια ερώτηση. Μας δώσατε διάφορα παραδείγματα για το που έχει γίνει η κατάχρηση τέτοιων τεχνολογίων και διάφορων εταιριών. Έχετε και παραδείγματα όπου οι εταιρείε έχουν πουλήσει τέτοιες τεχνολογίες σε μη κρατικούς φορείς, για παράδειγμα νομίζω ήταν το 2011, αν δεν κάνω λάθος, ή το 2012, δεν είμαι σίγουρη, όταν δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μια εταιρεία, μάλλον τηλεφωνήθηκα με μια εταιρεία η οποία έχει βάση στη Βαβαρία, η οποία συντηρούσε ε, εξοπλισμό στο Υπουργείο Εσωτερικών στη Συρία. Ήταν δύσκολο να πετύχω το τηλεφώνημα αυτό. Αλλά τους ε, ρώτησα, μάλλον μιας και δεν νοιάζει, δεν νοιαζόμαστε. Συγγνώμη. Ρώτησα λοιπόν τον εκπρόσωπο τη Γερμανική Εταιρεία Μέτρα στη Βαυαρία. Μια και δεν σα νοιάζει σε ποιον πουλάτε, θα μπορούσατε να πουλήσετε τα προϊόντα αυτά και στου αντιφρονούντε για παράδειγμα στη Συρία. Και η απάντηση ήταν θετική, γιατί όχι. Thank you very much. Σα ευχαριστώ. Η κυρία Κούστη Δύσκολο το όνομά σα. Δεν είμαι υπεύθυνη για το όνομά μου, ζητώ συγγνώμη. Τι να σας πω, ο πατέρας μου και ο παππούς μου ευθύνονται, αυτοί μου το έδωσαν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία το είπατε όμως. Σας ευχαριστώ όλους σας που ήρθατε εδώ σήμερα. Αυτό που μου κάνει εντύπωση κάπως είναι το γεγονός ότι στον τίτλο αυτό, με τον τίτλο αυτό, αν σωστά κατάλαβα, ε, επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στον, στους ελέγχους εξαγωγών. Λες και αν ελέγξουμε όλες τις εξαγωγές, όλες οι τεχνολογίες για την παρακολούθηση δεν θα υπάρχουν πλέον. Θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός στον κόσμο και ανταγωνιστικές εταιρείε που παράγουν τέτοια προϊόντα. Καλός και φανταστικός ο έλεγχος εξαγωγών λέτε. Σας πιστεύω. Παρ' όλα αυτά, αν ξέρουμε προς τα που εξαγάγονται τα προϊόντα, ξέρουμε και τι μπορεί να συμβεί, ποιος τι και ενδεχομένως μπορεί να ασκήσει κανείς έλεγχο. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε να περιοριστούμε απλά μόνο στο γεγονός ότι υπάρχει σύγχρονη τεχνολογία, την οποία όμως θα εξαγάγουμε. Οι εξαγωγές σχετίζονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα και γι' αυτό λοιπόν δεν καταλαβαίνω την κατηγορία. Το γεγονός ότι κατανοούμε και καταλαβαίνουμε ότι απότερη τμήμα της πολιτικής εξωτερικών υποθέσεων πλέον αποδεικνύει ότι η συγκήτρια κυρία Σάκη και εγώ Είμαστε πλήρη μέλη σήμερα στην Επιτροπή Διεθνού Εμπορίου και είμαστε παράλληλα πρακτικά μέλη και εδώ, στην Επιτροπή. Ακριβώ γιατί όλο και πιο πολύ επικρατεί η άποψη ότι και οι δύο τομεί δεν μπορούν πλέον να διαχωριστούν. Να θέσω το εξή ερώτημα προς όλου τους ομιλητέ. Πέρα από τον έλεγχο εξαγωγών. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πού μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, σε ποιους τομείς μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και να επηρεάσουμε τα πολιταρχικά καθεστώτα και τα άλλα κράτη. Σε σχέση με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών με έναν τρόπο που να συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τελευταία παρατηρήση, κάπω ε, ηρωνική κυρία Μιχάλσκι, μια και λέτε ότι θα πρέπει να είμαστε επικριτικοί για του προηγουλαλήσαντε. Πόσο κριτικοί, επικριτικοί είσαστε στις, στην ίδια σας την παρέμβαση. Έχετε και εκεί κάποιο σκεπτικισμό να μας αναφέρει Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριο Βασίλη. Κυρία Πρόεδρε, ούτε κι εγώ είμαι υπεύθυνο για το όνομά μου. Ο πατέρας μου μου το έδωσε. Είμαι υπερήφανο για το όνομά μου και ονομάζομαι Μπασίρ. Είναι μάλιστα ένα από τα ονόματα που ε, έδωσε, ε, που δόθηκαν στον προφήτη ε, Μωάμεθ και, και σημαίνει ο αγγελιοφόρος καλών ειδήσεων. Στην Αγγλία, στο Μάντσεστερ γεννήθηκα και θέλω να ε, ε, προσπάθησα να ε, ταξιδέψω χρησιμοποιώντας αυτό το σκάνερ το οποίο υπάρχει αλλά τελικά δεν έγινα αποδεκτός ε, προφανώς διότι αυτό το όνομα Μπασίρ δεν άρεσε στο μηχάνημα. Υπάρχουν βέβαια εκατομμύρια Μπασίρ αλλά προφανώς δεν ε, με άφησε να περάσω και φαντάζομαι ότι αυτό είναι αποτέλεσμα ε, του μαζικού προφάιλινγκ και της ε, μαζικής παρακολούθησης Βεβαίω κατανοώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην Ευρώπη όσον αφορά την τρομοκρατία και την αντιτρομοκρατική παρακολούθηση. Βεβαίω δεν το αμφισβητώ γιατί θέλω και εγώ ασφάλεια, αλλά παρόλα αυτά λέω ότι ε, δεν είναι δυνατόν να κάνουμε μαζική παρακολούθηση και μαζικό profiling του κόσμου. Πρέπει να είναι ε, στοχευμένο. Ε, εγώ επισκέφθηκα το Πακιστάν ε, εκεί όπου ε, εμψυχρό και σκοτώθηκαν, δολοφονήθηκαν εκατοντάδες άνθρωποι, κυρίως παιδιά, μετά από τρομοκρατική επίθεση των Ταλιμπάν. Βάσει παρακολούθησης και στοιχείων της παρακολούθησης η πακιστανική κυβέρνηση ε, κατόρθωσε να ε, καταλήξει ε, στο ποιοι ήταν αυτοί οι Ταλιμπάν οι οποίοι οδηγούμενοι από το Αφγανιστάν έκαναν αυτήν την τρομοκρατική επίθεση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είναι θετική η παρακολούθηση αλλά μετά πήγε και στο Χαράτσι όπου ε, ε, μου αναφέρθηκε ότι είναι δεκάδες ε, άνθρωποι οι οποίοι εξαφανίστηκαν ξαφνικά γιατί τους συνέλαβαν οι αστυνομικές αρχές. Δύο χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει που βρίσκονται ή τι κάνουν. Οι σύζυγοί τους, οι κόρες τους, τα παιδιά τους δεν ξέρουν που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν πολλοί αγνοούμενοι μεταξύ των οποίων πολλοί έχουν ήδη δολοφονηθεί. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να το δεχτούμε, είναι απίστευτο και ε, σκληρό. Ε, επομένως, μια ερώτηση στον κύριο Πέιτς μάλλον. Είπα ότι υπάρχει ένα θετικό στοιχείο της παρακολούθησης ε, γιατί επέτρεψε ε, στην κυβέρνηση να ε, βρει τα ίχνη των τρομοκρατών. Αλλά η ίδια κυβέρνηση χρησιμοποίησε μέσω των αστυνομικών δυνάμεων, των δυνάμεων ασφαλείας, αρνητικά την παρακολούθηση. Ε, επομένως, πώς είναι δυνατόν να ελέγξουμε τη χρήση, γιατί αυτό είναι το σημαντικό ερώτημα. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Φερνάδες Δεκοτέρο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και μετά, και μετά θα πάρουν το λόγο πολύ σύντομα όλοι οι πανελίστες. Δεκότ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φιλοξενεί μια τόσο σημαντική ακρόαση όπως είναι οι επιπτώσεις της ψηφιακής παρακολούθησης και των συστημάτων παρίστησης στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ελεύθερη κυκλοφορία online και offline είναι τμήμα της ε, δράσης μας τα τελευταία τρία χρόνια. Ως μέρος του σχεδίου αυτού, ήδη από το Μάιο του 2014, οι κατευθύνσεις αμέσως για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ελευθερία έκφρασης online και offline εγκρίθηκαν από τους Υπουργούς Εξωτερικών Υποθέσεων. Εδώ πολλοί Σύντομα θα ήθελα να περάσω σε κάποιες αρχές που αναφέρονται στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές και που έχουν άμεση σχέση με το δικό σας έργο. Η πρώτη είναι το δικαίωμα στην ελευθερία έκφραση, στον ιδιωτικό βία και στην προστασία των προσωπικών δεδομένων που μπορεί να παραβιάζονται εφόσον υπάρχει παρακολούθηση και υποκλοπές ή συλλογή προσωπικών δεδομένων, ιδιαίτερα όταν γίνονται σε μαζική κλίμακα. Ε, κάθε κράτος πρέπει να διασφαλίζει ότι ό,τι μέτρα λαμβάνονται για να προστατεύονται πληροφορίες αν συλλέγονται για την κρατική ασφάλεια πρέπει να συνάδουν με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει δεσμευτεί να προωθήσει μέτρα για την προστασία του ιδιωτικού βίου μεταξύ άλλων ζητώντας και από τρίτες χώρες να ευθυγραμμίσουν τη δικιά τους νομοθεσία σε ό,τι αφορά την διαφάνεια και να την προσαρμόσουν με το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Επίσης έχουμε δεσμευτεί να προωθήσουμε την καλή αυτή πρακτική και να διασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία που υπάρχει στις διάφορες χώρες όταν πρόκειται για παρακολούθηση, υποκλοπές και συλλογή προσωπικών στοιχείων να συμμορφώνεται προς τον νόμο και να τα αποκρίνεται πάντα με το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Θέλω τώρα να αναφέρω κάποιε πρόσφατε δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που εγκρίθηκαν οι κατευθυντήριε γραμμέ. Το πρώτο είναι ότι με του 18 διμερεί διαλόγου με διάφορε χώρε για την έγκριση των κατευθυντήριων γραμμών, εμεί υπογράψαμε το θέμα τη ε, έγκριση των νέων αυτών κατευθυντήριων γραμμών και ζητήσαμε από τρίτε χώρε να αναλάβουν αντίστοιχα βήματα. Επίση, Έχουμε και διαλόγου για τον κυβερνοχώρο με διάφορε χώρε όπου και εκεί ζητάμε την προστασία online των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί ενεργά προκειμένου να ενισχύσει τι προσπάθειε που γίνονται σε διεθνέ επίπεδα για την ελευθερία έκφραση online. Έχουμε προχωρήσει σε αποφάσεις επίσης όσον αφορά την προστασία του ιδιωτικού βίου. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεσμεύεται στην ε, συζήτηση που γίνεται σε διάφορα φόρα για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και θα συμμετάχουμε και στο Παγκόσμιο Φόρουμ. Προσβλέπουμε στη διάσκεψη της Χάγης που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο, όπου ελπίζουμε να προωθήσουμε την προοπτική αυτή της προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ψηφιακή σφαίρα. Συμμετέχουμε επίσης στο Διεθνές Δίκτυο και έχουμε εγκρίνει δήλωση βάσει της οποίας οι αρχές της διακυβέρνησης του δικτύου ε, πρέπει να περιλαμβάνει την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη ελευθερία έκφρασης, την προστασία του ιδιωτικού βίου και όλα αυτά πρέπει να διέπουν τη διακυβέρνηση του διαδικτύου και να ισχύουν online. Τώρα δουλεύουμε πάνω στα συμπεράσματα της διπλωματίας ε, για τον κυβερνοχώρο μέσα σε μια ομάδα εργασίας. Έχουμε μια συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο διαδίκτυο και αναγνωρίζουμε ότι οι αξίες αυτές θα συνεισφέρουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη προκειμένου να προστατεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, ε, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για τα συμπεράσματα που δημοσιεύτηκαν το 2014 όσον αφορά όλου του τομείς του κυβερνοχώρου. Έχουμε δημιουργήσει και μία άτυπη εσωτερική υπηρεσία για το θέμα αυτό που ασχολείται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει το έργο της και μέσα στο 2015. Διάφορα συμβάντα είχαμε και σε διάφορα γεγονότα προσπαθήσαμε να υπογραμμίσουμε τη σημασία που έχουν όλα αυτά. Τον Μάρτιο, για παράδειγμα, υπήρχε μια συνάντηση του ΟΑΣΕ επ' αυτού. Και ένα από τα σημαντικά θέματα που τέθηκαν εκεί και που πρέπει να προσέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τις παράνομες υποκλοπές και επίσης πρέπει να ξέρετε ότι προσφέρουμε και κατάρτιση σε αξιωματούχους των χωρών μελών όσον αφορά τη σχέση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την παρακολούθηση και τις υποκλοπές και την προστασία του προσωπικού βίου. Το 2014 είχαμε και ένα πάνελ με ενημέρωση και πάλι πάντα για την ισορροπία ανάμεσα στην παρακολούθηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για να ολοκληρώσω, επιτρέψτε μου να σας πω και το εξής. Η Ευρωπαϊκή Πίεση Εξωτερικής Δράσης δουλεύει αυτή την εποχή σε ένα πρόγραμμα δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, χρησιμοποιώντα την εμπειρία της από τα διάφορα αυτά γεγονότα, διάφορες διασκέψεις που έγιναν ε, πρόσφατα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, δύο λεπτά ο καθένας να απαντήσουν οι προσκεκλημένοι μας και τέλος η συγκεκριά μας. Αρχίζουμε από τον κύριο Λαρίου παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Δύο πολύ σύντομα σχόλια. Η πρώτη ερώτηση ρωτούσε ποια είναι η συγκεκριμένη διασύνδεση ανάμεσα στην ε, τεχνολογία και την εξαγωγή τεχνολογίας και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι σε σχέση με τα κράτη μόνο. Ε, νομίζω ότι το πρώτο είναι ότι πρέπει να πούμε ότι όλες ε, οι χώρες, όλες οι κυβερνήσεις οφείλουν να οδηγηθούν προς την ανάπτυξη και μέσω εξαγωγών ε, αλλά οπωσδήποτε μέσα στα πλαίσια της πλήρους προστασίας των δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα στα πλαίσια όμως της καθολικότητας των των ε, αρχών ε, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, υπάρχει και η υποχρέωση της προστασίας των δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον πλανήτη και όχι μόνο στη συγκεκριμένη χώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν μιλάμε για αδειοδοτήσεις εξαγωγών άλλωστε. Δεύτερον, υπάρχει και ένα στοιχείο εταιρική κατά κάποιο τρόπο ε, ευθύνη. Ε, δεν θα μπω ε, σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά έχουμε μια σχετική έκθεση με εισηγητή τον Ζαν Ρόκι που αφορά ακριβώς αυτήν την εταιρική ευθύνη ευθύνη ε, μια και το κάθε τμήμα της ε, κοινωνίας έχει ε, μια υποχρέωση, ένα κομμάτι υποχρέωσης και οι όμιλοι, οι εταιρείες επίσης έχουν μια υποχρέωση. Οι ίδιες οι εταιρείες, λοιπόν οι ίδιοι οι όμιλοι θα πρέπει να καταλάβουν σε ποιους ακριβώς πουλάνε την τεχνολογία τους. Τέλος, να πω το εξής. Ε, κανείς ε, δεν σχολίασε τι σημαίνει για μας, για τον καθένα χωριστά. Αυτό όμως είναι μια πάρα πολύ σημαντική σκέψη. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο χωρίς ε, να ε, δούμε τι ε, εμείς κάνουμε γι' αυτό. Δεν μπορεί να είμαστε μέλη, μέρη ενός κράτους ή μιας κοινωνίας που αναπτύσσει σύμφωνα με το δίκαιό της <clears throat> τεχνολογίες οι οποίες όμως χρησιμοποιούνται για την κατάλυση δικαιωμάτων σε άλλες ε, ε, ε, πλευρές του κόσμου, σε άλλα σημεία του κόσμου. Γιατί εν τέλει κινδυνεύουμε και εμείς οι ίδιοι από αυτήν την κατάλυση των ε, δικαιωμάτων. Επομένως, ναι, επιτήρηση στα πλαίσια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μονάχα οι ισχυρές δημοκρατίες μπορεί να έχουν σωστή, ισχυρή επιτήρηση για να έχουν και ισχυρή ασφάλεια. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για τι ερωτήσει που μου κάνατε. Θα ήθελα να τι απαντήσω και τις δύο. Και την ερώτηση τη κυρία Λοχπίλερ και της κυρίας Νορού με το ερώτημα που έχει μόχλευση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα. Και το ερώτημά σας για την χρήση των τεχνολογιών με τρόπο που να συνάδει με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εγώ πιστεύω ότι επικεντρωθήκαμε ίσω υπερβολικά στην εξαγωγή των τεχνολογιών εξαγωγών ε, παρακολούθησης. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι σημαντικό αυτό, είναι σίγουρα ένα πολύ κεντρικό σημείο. Αλλά είναι σωστό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στραφεί προς αυτό το συνδυασμό εμπόριο και ανθρώπινα δικαιώματα και να ασχοληθεί πιο επισταμένα με το θέμα αυτό και έτσι να μην επικεντρωθούμε μόνο στις ε, ελέγχους εξαγωγών ή να μην έχουμε την ψευδέστηση ότι μόνο με ελέγχους εξαγωγών θα επιλύσουμε το πρόβλημα. Μπορούμε να καταρτήσουμε καταλόημα και μπορεί να γίνει διαφοροποίηση σωστή με τον τρόπο αυτό, αλλά εκεί όπου βλέπω ότι υπάρχει μόχλευση και δυνατότητα μόχλευση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσω και καθήκον μόχλευση με επιλεκτικό τρόπο να πω, είναι το εξή. Δεν είμαστε μόνο εξαγωγή προϊόντων και τεχνολογιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται εξαγωγέας και προτύπων για τη δημοκρατία, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ως τέτοιος εξαγωγέας θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα μόχλευσης. Δεν θα είναι τόσο μεγάλη η μόχλευση ενδεχομένω σε χώρες όπως η Κίνα ή το Ιράν. Αυτό θα ήταν πραγματικά μη ρεαλιστικό να μην το αναγνωρίσουμε. Αλλά εκεί που έχει μόχλευση η Ευρωπαϊκή Ένωση, στη γειτονιά της για παράδειγμα και κύριε Βάιτχολτερ, ή στο πιο νέο περιβάλλον, στην πολιτική γειτονία, εκεί θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντω μπορεί με τις δυνατότητες που έχει στα χέρια της, όχι μόνο με τον έλεγχο των εξαγωγών, αλλά και με τη σύνδεση με άλλες, για παράδειγμα, εμπορικές σχέσεις Εκεί μπορεί να έχει αντίκτυπο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να κοιτάξουμε μόνο το τεχνολογικό σκέλος, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθούμε και σε ερωτήματα του πώς μπορεί η ψηφιακή τεχνολογία στα πλαίσια της κοινωνίας των πολιτών και των συμφερόντων των διάφορων ομάδων. Πώς μπορεί λοιπόν να προωθηθεί και να ενισχυθεί αυτή η πτυχή. Να υποτίξω το εξή. Κοιτώντα τη σχέση που υπάρχει μεταξύ διείσδυση του διαδικτύου στι χώρε και το βαθμό τη ελευθερία του διαδικτύου, κοιτώντα λοιπόν ποιο είναι ο συσχετισμό των δύο ε, στοιχείων καταλήγουμε σε μια ομάδα χωρών όπου υπάρχει μεγάλη ελευθερία ανάπτυξης. Μια ομάδα χωρών όπου αν αναπτυχθεί κι άλλο η τεχνολογία με τους κοινωνικο-οικονομικούς όρους που συνδέονται φυσικά με την αναπτύξη αυτή είναι ανοιχτό κατά πόσον αυτές οι χώρες θα κινηθούν πιο πολύ προς τη δημοκρατική οδό ή πιο πολύ, πιο πολύ προς την ε, κατεύθυνση του, της λογοκρισίας της υψηλής τεχνολογίας. Εκεί ναι. λοιπόν μπορούμε να ασκήσουμε επιρροή. Αν επικεντρωθούμε πιο πολύ στις χώρες αυτές, νομίζω ότι θα έχουμε εντοπίσει ε, μια σημαντική ομάδα χωρών όπου μπορούμε να έχουμε ουσιαστικό αντίκτυπο. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Page. Ευχαριστώ. Για την κυρία Λόκεμπερτ. Για τους μη κρατικούς ένα πράγμα θα το σταματούσε αυτό ανεξαρτάται από την ίδια την επιχείρηση αν νιώσει ότι δεν είναι υποχρεωμένη να πουλήσει. Τα τεχνικά στοιχεία κάποιων τεχνολογιών σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στην επικοινωνία. Μόνο οι φορείς που έχουν πρόσβαση, που είναι κυβερνητικοί, συνήθως μπορούν να κάνουν κάτι. Όσοι χρησιμοποιούν λογισμικό παρίστησης, τεχνικά τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει την πώληση και την αγορά τέτοιου λογισμικού. Είναι πολύ πλούσιοι ιδιώτες που θέλουν να το χρησιμοποιούν. Ξέρουμε και σχόλια από διάφορες επιχειρήσεις. Μια Ιταλική πρόσφατα είπε ότι είμαστε προσεκτικοί που πουλάμε, δεν πουλάμε όπου να είναι. Παρ' όλα αυτά φτάνει τέτοιο λογισμικό σε χώρες όπως το Καζαχστάν, Σομαλία. Γι' αυτό που είπε ο κύριος Βασίρ. Ναι, υπάρχει θεμητή τέτοια πώληση, εξαρτάται σε ποιο καθεστώς. Μπορείς να πουλήσεις τεχνολογία και μετά να ελέγξεις τη χρήση της. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Το βλέπουμε με την τεχνολογία την αγγλική και τη γερμανική που έχει πουληθεί στο Μπαχρέιν. Μετά τη χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν κόσμο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έτσι κι αλλιώ το Μπαχρέιν δεν υποσχέθηκε ποτέ ότι θα χρησιμοποιεί την τεχνολογία αυτή μόνο στην χώρα. Χρησιμοποιείται και σε άλλες χώρες. Δεν μπορείς να το σταματήσεις αυτό στα σύνορα. Την κυρία Ρόβαλ θέλω να πω ότι η εξαγωγή τεχνολογίας διευκολύνει την καταστολή στο Τουρκμενιστάν, για παράδειγμα, 190 97 στις 198 χώρες, έχει την 127η θέση ε, όσον αφορά την ε, καταπίεση των ελευθεριών. Και όμως, η τελική χρήση και ο τελικός ε, χρήστης όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το ζητούμενο. Και πρέπει να το ψάχνουμε πριν προχωρήσουμε σε εξαγωγές. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Όσον αφορά το θέμα που μας ε, απασχολεί και για την αύξηση της ε, ψηφιακής ασφάλειας νομίζω ότι πλέον ε, οι πρωταγωνιστές της ε, των τεχνολογιών ε, ε, της, της κοινωνίας των πολιτών συγγνώμη, ζητούν και απαιτούν όλο και περισσότερο ασφαλή τεχνολογία. Το σημαντικό το οποίο πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι η στήριξη της, την εκπαίδευση και της προσπάθειες ασφάλειας θα πρέπει να είναι μακροχρόνια και όχι μια και γιατί η συζήτηση για την ασφάλεια είναι η ιδιαίτερα περίπλοκη, προϋποθέτει και γνώσεις ε, και ε, εμπειρία και επομένως θα πρέπει να είναι πάντα μακρόθωρη και οπωσδήποτε να γίνεται ε, με στήριξη και της κοινωνίας των πολιτών και των ακτιβιστών και τα λοιπά, έτσι ώστε να αυξηθεί η συνειδητοποίηση και να γίνεται και βάση όσο γίνεται περισσότερο της χρήσης των πλατφορμών επικοινωνίας. Τώρα, ε, πώς είναι δυνατόν να ελέγχουμε τις, ε, τους εξοπλισμούς ε, τους οποίους πουλάμε σε άλλες χώρες. Νομίζω ότι ένα πρώτο βήμα είναι να ξεκινήσει διάλογος με τις εταιρείες σχετικά με το τι είναι δυνατόν και τι πρέπει να απαιτηθεί από αυτές. Ε, γιατί πολλές φορές ε, υπάρχουν ε, συμβόλαια, γίνονται συμβόλαια ή παρέχονται υπηρεσίες από αυτές τις εταιρείες και επομένως θα πρέπει να ξέρουμε τι είναι δυνατόν να κάνουν οι εταιρείες αυτές σε σχέση με τους πελάτες τους, τι μπορούμε να απαιτήσουμε, τι μπορούν να δώσουν εκείνου, ποιες είναι οι απαιτήσει που θα πρέπει να έχουμε όσον αφορά την λογοδοσία και την τακτική αναφορά από αυτές τις εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mrs. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μακίνα. Ο κύριος Μισάλσκι. Θα είμαι σύντομος. Για το ερώτημα του κατά πόσον υπάρχει εναλλακτική για τους ε, ελέγχους εξαγωγός. Ευτυχώς οι οδηγίες και τα γραμμές είναι μόνο κατευθυντήρες γραμμές, δεν είναι ακόμα δεσμευτικές. Ε, δεν είναι το πιο επιτιδευμένο και το πιο κομψό μέτρο, αν θέλετε, η έλεγχη εξαγωγών, αλλά είναι το πιο αποτελεσματικό και θα πρέπει ω οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων να είμαστε ρεαλιστέ και να δούμε πώ μπορούμε πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά να εξωτεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, του ανθρώπου. Αυτό είναι ο μοναδικό τρόπο αποτελεσματικό τον οποίο θεωρούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή για να αποτρέψουμε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κατά πόσον ε, έχω και εγώ κριτική να ασκήσω στον εαυτό μου, όπω ε, και στον κύριο Φοκούμη. Σε κάποιε περιπτώσει ναι, να σα πω την αλήθεια. Α, φυσικά και πάντα θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι να κάνουμε αυτοκριτική για αυτά που κάνουμε σε σχέση με όλους τους άλλου παράγοντε, σε όλου του τομείς. Και εδώ θα επανέλθω σε αυτά που είπαμε στην αρχή. Δυστυχώς ε, η έλεγχη εξαγωγών αυτή τη στιγμή είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο. Ο κ. Μασίρ ανέφερε κάτι το οποίο αποτελεί πολύ ακαθόδε ζήτημα. Από τη μία έχουμε την νόμιμη παρακολούθηση τουριστών, εγκληματιών. Από την άλλη έχουμε και την κατάχρηση της παρακολούθησης αυτής σε χώρες όπου δεν είναι σαφή τα σύνορα, τα όρια θα πρέπει να ελέγχουμε, να απαγορεύσουμε ενδεχομένω την εξαγωγή τέτοιων προϊόντων. Το θέμα είναι κατά πόσο οι μυστικέ υπηρεσίε του παρακολουθούν και τους Ταλιμπάν με τις ε, τεχνολογίες παρακολούθησης ή αν απλά αποδίεται στην παλιά καλή κατοσκοπία. Γιατί νομίζω ότι και σε ό,τι αφορά τους Ταλιμπάν δραστηριοποιείται. Sí, voy a dar un minuto la palabra, bueno, un minuto no, medio. Ενάμιση λεπτό στον κύριο Λαρίου. Τρία δευτερόλεπτα. Ξέχασα να πω ότι οι αρχές και οι guidelines ε, μου που έχουν ε, οριστεί μου φαίνονται εξαιρετικό πρώτο βήμα. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όλες οι πολιτικές τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, μεταξύ των οποίων και η ρύθμιση των εξαγωγών να ε, είναι ε, να συνάδουν με αυτές ε, τις guidelines. Ναι, πραγματικά είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Η Excellent... Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσω και όλους σας για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις και που μείνετε μαζί μας αυτή τη μακρά ακρόαση. Ακούσαμε πολλές προτάσεις και μια εντελεχή ανάλυση της κατάστασης όπως εξελίσσεται. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι η ασφάλεια και τα εμπορικά συμφέροντα και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν πρέπει να είναι αυτοαναιρούμενα. Θα πρέπει να συνάδουν τα μεν με τα δεν. Πρόκειται για μια αγορά πολλών εκατομμυρίων με αδιαφάνεια και με μεγάλου κινδύνου. Αλλά οι κίνδυνοι για την ασφάλειά μα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα του κόσμου σε όλο τον κόσμο είναι τόσο σημαντικά που δεν μπορούν να μα οδηγήσουν να αποδεχθούμε το status quo της, ε, του νομικού κοινού που υφίσταται. Θα πρέπει να καλυφθεί αυτό το χάσμα. Φυσικά δεν είναι πρόθεσή μας να εμποδίσουμε την έρευνα, δεν είναι ε, πρόθεσή μας να αναλυθούμε σε πολέμους κρυπτογράφησης. Έχουμε μάθει το πάθημά μας, από τα πάθηματά μας. Να δούμε λοιπόν ε, που έχουμε ευαισθησία. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πουλάμε αυτή την ευαλωτότητα σε καθεστώτα απολυταρχικά και επικίνδυνα. Θα ήθελα να απευθύνω μία ανοιχτή πρόσκληση στο Φουκάμι και στους άλλους εμπρεγνώμονες στο Kale Computer Lab να συνεργαστούν μαζί μας προκειμένου να καταλήξουμε σε ευφύη ευρωπαϊκή νομοθεσία όπου θα αντιμετωπίζουμε με σωστό τρόπο όλε τι ανησυχίε, αλλά θα ληφθούν υπόψη και τα συμφέροντα τη τεχνολογία εχμή. Χρειαζόμαστε ευφυείς πολιτικέ, θα πρέπει να είμαστε πιο ακριβεί από αυτά που συμφωνήθηκαν στο Βάσεναρ. Και θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να είναι πιο υψηλός ο πύχης. Να μην θεωρήσουμε λοιπόν ότι είναι μοναδική λύση αυτή που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πραγματικά να δημιουργηθεί μια αρχή για να καταρτήσουμε ευφύ νομοθεσία. Και όσοι είπαν ότι η αυτορύθμιση θα μπορούσε να αποτελέσει λύση. Ας το ξανασκεφτούν γιατί υπάρχουν διάφορες επιχειρήσεις στην αγορά αυτή που έχουν ε, ένα δημόσιο όνομα αλλά να σας, ε, να σας διαβεβαιώσω ότι οι πιο μεγάλοι φορείς ε, δρούν στο σκοτάδι, δεν έχουν κάποιο όνομα να χάσουν. Δεν προβάλλονται στη δημοσιότητα. Δεν είναι λοιπόν αυτό λύση για όλη την αγορά. Και είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι η συζήτηση αυτή θα πρέπει να αποτυπώνει και τις ε, χώρες και τις ευρωπαϊκές πολιτικές, αλλά η αρχή που εξέφρασε ο κ. Λαρού ότι η μαζική παρακολούθηση είναι πάντα αντίθετη με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σημαντική. Θα πρέπει να αποτελέσει σημείο αφετηρία. Και φυσικά έχουμε και πρότυπα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, πρότυπα που θέτουμε εμεί εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έτσι απαντώ και στη συναδελφή Χοντελήφε. Γιατί εμείς θέτουμε λοιπόν πρότυπα για το πώς θα μορφώνονται τα συστήματα τηλεπικοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προαπαιτεί τα δίκτυα, για παράδειγμα τηλεπικοινωνίας, να έχουν μια νόμιμη οδό α, υποκλοπών σε περίπτωση που η αστυνομία νόμιμα θέλει να κάνει μετά από εισαγγελική εντολή έρευνα σε περίπτωση τρομοκρατίας. Λοιπόν, έχει σημασία ποιος αποφασίζει το ότι είναι νόμιμο και τι όχι. Αν δούμε τα πρότυπα αυτά στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, το οποίο τόσο πολύ θέλουμε να προστατεύσουμε στην Ευρώπη, έχει μεγάλη διαφορά να εξαγάγουμε αυτά τα συστήματα σε χώρες όπου έχουμε επανειλημμένα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κρά... κράτος δικαίου και έτσι ανοίγουμε την πίσω πόρτα σε κλιματικέ δραστηριότητε, σε κατασκοπία κατά των πολιτών, των ακτιβιστών, σε οποιονδήποτε, κατά οποιοδήποτε ανθρώπων που ενδεχομένω να γίνονται αντιληπτήρε επικίνδυνοι. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε το τι πολλούμε και πού το πολλούμε και τι συμβαίνει στις χώρες αυτές. Έχουμε τόσες περιπτώσεις όπου υπήρξε ανοιχτή καταγγελία από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση διαφόρων καθεστώτων, αλλά δεν αναρωτιόμαστε με τι εργαλεία λειτουργούν αυτά τα καθεστώτα και κατά πόσον τα εργαλεία αυτά έχουν κατασκευαστεί στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να αποτρέψουμε τέτοιες τεχνολογίες που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιούνται για κατασταλτικά μέτρα. Και ήμουν περίεργη να μάθω τι θα περιλαμβάνει αυτό το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αραβικού Συνδέσμου. Γιατί αφενός έχουμε καλές κατευθυντερίες γραμμές, τις οποίες χρησιμοποιεί η υπηρεσία εξωτερικής δράσης για τα θέματα online-offline, αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι γίνονται διαγωνισμοί από την Αιγυπτιακή κυβέρνηση για ευρωπαϊκή τεχνολογία η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την καταστολή. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο και μάλιστα κατεπίγουσα ανάγκη για να καταρτιστεί μια φιλόδοξη ατζέντα για τα επόμενα βήματα. Θα πρέπει να είναι η ηγετική φυσιογνωμία η Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένως αυτό να είναι δύσκολο για τα συμφέροντα της αγοράς, αλλά νομίζω ότι διακυβεύεται κάτι πολύ πιο σημαντικό. Η ευθύνη μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο παγκόσμιο προσκήνιο. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική προσέγγιση και γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι τόσο σημαντική αυτή η ακρόαση για να δούμε πώς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το εμπόριο αλληλεπηρεάζονται σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα της τόσο ταχείας αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να νιώθετε ότι η ακρόαση αυτή σας βοήθησε να συντάξετε την έκθεσή σας, που θα είναι σίγουρα ξέρετε. Τέλος. Και πέρα από το γεγονό ότι η Γενική Διεύθυνση Connect δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα, γιατί είχαν ε, μια σημαντική εκδήλωση ούτε και η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και η ΔΕΦΚΟ δεν το θεώρησε απαραίτητο να έρθει. Παρ' αυτά, είναι μαζί μας ο κύριος Πάολο Αρζότη από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε εδώ και σας δίνω το λόγο ευθύ αμέσω. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά πώς είναι δυνατόν με τόσο κόσμο που έχετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην βρήκε κανείς το χρόνο μια τόσο σημαντική μέρα σαν τη σημερινή να έρθει εδώ στην Υποπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εσείς όμως παραμείνατε εδώ όλο το πρωί και έτσι ευχαρίστω σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, είμαστε εδώ και παραμείναμε εδώ γιατί είναι θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Είμαστε και εμείς σε διαδικασία μεταρρύθμισης. Η πρώτη προφορική ερώτηση που απαντήθηκε είναι σχετική. Τα ανθρώπινα δικαιώματα εμείς τα βάζουμε σαν προϋπόθεση. Ε, δεν κάνουμε εξαγωγές εφόσον δεν τηρούνται αυτά. Θέλω να απαντήσω στην κυρία Λοχμπίλερ όμως. Η έλεγχη εξαγωγών αποτελεί ένα μέσο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Αν γνωρίζουμε ότι ένα κράτος δεν έχει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη χρήση της τεχνολογίας, έχουμε και άλλα μέσα. Έχουμε τις κυρώσεις, άρθρο 15 της συνθήκης, και μπορούμε επίσης να κοιτάξουμε και το ευρύτερο πλαίσιο των εργαλείων που έχει στη διάθεσή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, για τη γενική μας διεύθυνση πρέπει να ξέρετε ότι βεβαίως και θέλουμε να είμαστε εδώ και να παρακολουθούμε τις συζητήσεις σας που είναι τόσο ενδιαφέρουσες. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έχουμε ήδη μαζί μας τον επόμενο προσκεκλημένο μας για να συζητήσουμε για τη Βόρεια Κορέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους όλους τους προσκεκλημένους για τις εξαίρετες παρουσιάσεις σας, παρόλο που είχατε λίγο χρόνο στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ.